Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλημέρα σε όλους σας. Καλωσορίσατε κύριε Dirk Άνερ στην Επιτροπή μας. Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής θα μας δώσει ε, μία έποψη της εκτέλεσης του προϋπολισμού 2009. Θα παρουσιάσει λοιπόν τις ε, πληρωμές, ε, τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές σχετικά με την τεχνική αρρωγή. Επίσης θα ασχοληθεί με το θέμα του του περιορισμού των αυτόματων δεσμεύσεων. Thank Σας δίνω το λόγο αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. δεν ε, φαντάστηκα ότι ε, θα ε, μπορούσα να σας κάνω μια εξαιρετική παρουσίαση με powerpoints και τα λοιπά. Αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και είπα ότι καλύτερα θα ήταν να έχουμε μια καλή συζήτηση για τα μεγάλα στοιχεία, τους μεγάλους αριθμούς, να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια προοπτική στην συζήτηση αυτή. Προτίμησα λοιπόν ε, να προετοιμάσω και ένα υπόμνημα με όλες τις πληροφορίες ε, για σας έτσι ώστε να τα έχετε έτοιμα ε, και να μην έχετε σήμερα τον προβληματισμό αυτό των υπερβολικών λεπτομεριών. Θα σας στείλουμε λοιπόν ένα σύντομο υπόμνημα σε μερικές μέρες και θα δείτε αναλυτικά όλα τα αριθμητικά στοιχεία. Μπορώ να είμαι και λίγο ε, υπερήφανος για την εκτέλεση του ε, προϋπολογισμού και όσον αφορά τις δεσμεύσεις και όσον αφορά τις ε, πληρωμές φτάσαμε στο 99,9% του προϋπολογισμού και στην πραγματικότητα όσον αφορά τις πληρωμές πρέπει να πω ότι στην ουσία ξεπεράσαμε ακόμα και αυτό το μεγάλο ποσοστό και θα σας εξηγήσω γιατί. Έχουμε Είχαμε λοιπόν ένα συνολικό ποσό πληρωμών για πέρσι και εδώ θέλω να με ελέγξει ο συνάδελφός μου, τον οποίον ο εξεβονίμων καθήμενα, τον οποίο θα ήθελα να σας τον παρουσιάσω μάλιστα και ο οποίος είναι επικεφαλής ε, των οικονομικών υπηρεσιών. Πληρωμές λοιπόν που έγιναν πέρσι 26 26,7 ε, δις ε, ευρώ. Εξ αυτών των 26,7 δις, 18,3 δις για το Περιφερειακό Ταμείο και 7,1 για το Ταμείο Συνοχής. 25,4 λοιπόν ε, περίπου, 26,7 σύνολο, 25,4 για το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνεχής. Τα υπόλοιπα είναι μικρότερα ποσά για το Ταμείο Αλληλεγγύης, την ΙΣΠΑ, καθώς και πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Ας δούμε τώρα από πιο κοντά αυτά τα 25,4 δις τα οποία ανέφερα προηγουμένως ε, για το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. 25,4 δις λοιπόν τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερο ε, από αυτό που είχαμε προβλέψει. Ε, δηλαδή είναι περίπου 105% ε, από τα αρχικώς προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό και καταφέραμε να κάνουμε τις πληρωμές αυτές γιατί κάναμε μία μετατόπιση πόρων από το Κοινωνικό Ταμείο στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το συνολικό ποσό των 25,4 το ενδιαφέρον σε αυτό το ποσό, τα 25,4, είναι αυτά τα 7 εκατομμύρια, τα οποία ακόμα ε, συνδέονται με την περίοδο 2000-2006 και 18,4 18,4 δις συνδέονται με το 2007-2013 με τη νέα περίοδο δηλαδή. Ας δούμε τώρα καλύτερα αυτά τα 18,4 δις τα οποία μόλις ανέφερα. 18,4 λοιπόν από το 2007-2013. 9 δις ακόμα ε, πρόκειται για προκαταβολές. Ε, θα θυμάστε ότι ε, σε σχέση με, το, ε, τα ποσά τα οποία δόθηκαν ε, για τη διάσωση των οικονομιών το 2008 είχαν δοθεί τα χρήματα αυτά για το σύνολο των, του κοινωνικού ταμείου και το, του Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης και επομένως ξεκινήσαμε με 8 περίπου εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια στην αρχή και μετά άλλα 11 δις 11 δις λοιπόν για τις ε, περίπου 9 δις ε, για το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Ε, επανέρχομαι τώρα. Πέρυσι είχαμε ήδη 9,4 δις ευρώ φρέσκο χρήμα τα σχετικά με περιπτώσεις που ζήτησαν χρήματα τα κράτη-μέλη και δώσαμε τα χρήματα αυτό. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μία απομείωση ε, και στον δικό μας προϋπολογισμό όσον αφορά τα προγράμματα 2007-2013. Και η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο προφανής αν δούμε τα χρήματα ε, και τις απαιτήσει που είχαμε περί τα τέλη του προηγούμενου χρόνου και που δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε γιατί τα περιθώρια ήταν πάρα πολύ στενά στα τέλη του προηγούμενου χρόνου ε, και οι επιστροφές θα γίνουν αρχές αυτού του χρόνου. Και φτάνουμε λοιπόν στα 6,2 περίπου δις Πέρσι λοιπόν όσον αφορά τη νέα περίοδο είχαμε 9 δις ε, προκαταβολές 9,4 ε, δις απαιτήσει μετεπιστροφών για την προηγούμενη χρονιά και υπολοιπόμενο 6,2 ε, δις απαιτήσει του προηγούμενου χρόνου αλλά επιστροφές αυτού του χρόνου που ήδη έχουν ξεκινήσει εντωμεταξύ οι επιστροφές αυτές, οι πληρωμές αυτές. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η κατάσταση που σας παρουσίασα ε, μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει καλά τα προγράμματα της νέας περίοδου και μπορώ να πω κύριε Πρόεδρε ότι, να πω λοιπόν ότι μέχρι ένα βαθμό πιστεύω ότι τελικά καταφέραμε να σεβαστούμε πλήρως τη σύμβαση την οποία είχαμε, ε, την υποχρέωση αν θέλετε την οποία είχαμε αναλάβει ε, στο, με το πακέτο στήριξης. Ε, δηλαδή ναι, κάναμε κάποιες πρώτες βαριές πληρωμές έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη ρευστότητα στα κράτη-μέλη και βεβαίως κάναμε και κάποιες λέτε από τη δική μα πλευρά για να δούμε αν χρησιμοποιήθηκε σωστά αυτή η ρευστότητα από τα κράτη-μέλη και μπορούμε να πούμε ότι ναι, για το έτος 2009, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες καταφέραμε να συλλέξουμε από τα κράτη-μέλη, ναι λοιπόν, τα κράτη ε, χρησιμοποίησαν ε, τα χρήματα ε, πρώτον για πρώτες πληρωμές, για προκαταβολές και σε μερικές περιπτώσεις σαν συμπλήρωμα της συγχρηματοδότησης. Αυτό όσον αφορά τα 9 δις από το Ταμείο ε, Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Επιπλέον όμως των 9 έχουμε και τις ενδιάμεσες πληρωμές. Για να γίνουν ε, οι ενδιάμεσες πληρωμές θα πρέπει να υπάρχει ένας λογαριασμός ο οποίος θα υποβληθεί, θα ε, ε ελεγχθεί και βεβαίως μετά ε, φτάνουν οι απαιτήσει στην Επιτροπή. Αυτό που είδαμε και είναι ενδιαφέρον να το αναφέρουμε είναι ότι στην ουσία, στην πράξη μάλλον, ε, η διαδικασία αυτή στην ουσία ξεκίνησε κανονικά το δεύτερο μισό του 2009. Υπήρχε η προπαρασκευαστική περίοδος 2007-2008 αλλά απογειώθηκε στην ουσία το τελευταίο κομμάτι του 2009 και η εξήγηση είναι απλή. Αυτό που συνέβη είναι ότι στα πλαίσια του πακέτου στήριξης ε, χρειάστηκε να επιμηκύνουμε ε, τις τελικές προθεσμίες πληρωμής για την περίοδο 2006 την επιμηκύναμε κατά 6 μήνες. Ευχαριστώ μέχρι τέλη Ιουνίου 2009 και στην ουσία αυτό που συνέβη είναι ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη, οι περισσότερες περιφέρειες εδράχθησαν τις ευκαιρίες ε, έτσι ώστε ε, να χρησιμοποιήσουν όσο γίνεται περισσότερο ε, τα χρήματα τα οποία ήταν ακόμα διαθέσιμα την περίοδο 2000-2006 και επομένως όλοι οι πόροι, όλοι, όλοι οι πόροι οι οποίοι παρέμεναν μεταφέρθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν από την περίοδο 2000-2006 ε, και κατά κάποιο τρόπο παρέμειναν στο ντουλάπι οι ε, πληρωμές του, του 2007-2013. Επομένως, στην ουσία, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δουλέψει ε, στο, για το 2000-2006 όταν τελείωσαν οι πληρωμές αυτές μετέφεραν την δραστηριότητά τους το 2007-2013 ε, και επομένως ε, και αυτό αφορούσε όλες τις διαδικασίες ε, πιστώσεις, πληρωμές, απαιτήσει κλπ. Αυτό ήταν η πρώτη μας υποχρέωση, δηλαδή να φέρουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ρευστότητα στα κράτη-μέλη μέσω των προκαταβολών. Και το δεύτερο σκέλος της υποχρέωσής μας ήταν ότι θα προσπαθούσαμε να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να τους ε, ε, πείσουμε να ξεκινήσουν την εφαρμογή των πολιτικών επιτόπου και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήδη είχαμε ε, καθυστέρηση, περίπου δωδεκάμινη καθυστέρηση, σε σχέση με τα φυσιολογικά όρια κατά την άποψή μας και δεύτερος λόγος και πιο σημαντικός ήταν η κρίση και το γεγονός ότι θέλαμε άμεσα και απόλυτα να ληφθούν μέτρα επιτόπου έτσι ώστε ε, να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά ε, την ζήτηση αφενός και από την άλλη πλευρά βεβαίως να γίνουν ε, οι απαραίτητες επενδύσεις γιατί πιστεύουμε ότι αυτού του είδους οι έξυπνες επενδύσεις, smart investments όπως τις ονομάζουμε, θα ήταν πολύ χρήσιμες για το μέλλον. Αυτό συνέβη λοιπόν σε ένα μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του έτους 2009 ε, και αυτό ε, ε, και ξεπεράστηκε ξεπεράστηκαν δύο μεγάλα προβλήματα τα οποία είχαμε. Το ένα μείζον πρόβλημα ήταν βεβαίως η ίδια η κρίση, η οποία σε ορισμένα κράτη-μέλη οδήγησε σε τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα και επομένως είχαν δυσκολία να βρουν το ποσοστό συνχρηματοδότησης ε, το οποίο είναι απαραίτητο για την πολιτική συνοχή και ε, επίσης πολλές χώρες ε, είχαν την άποψη ότι ναι θα κάνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη αποταμίευση αλλά το τελευταίο που μας ενδιαφέρει είναι στην ουσία αυτό το σκέλος της διαρθρωτικής πολιτικής μέσα από το Ταμείο Συνοχής. Εν πάση περιπτώσει όμως υπήρχαν και κάποιες ε, χώρες μέλη, λίγες, ε, οι οποίες έδωσαν την εντύπωση ότι η κρίση πραγματικά συνέθλιψε την ε, ικανότητα εθνικής συγχρηματοδότησης και επιπροσθέτως να πούμε ότι ε, μέχρι πέρσι πολλές ε, χώρες μπορούσαν να, ε, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τις προκαταβολές για να κάνουν αυτή την εθνική συνχρηματοδότηση. Αντιθέτως, σε μια-δυο περιπτώσεις είδαμε ε, το πρόβλημα των εθνικών αντικυκλικών προγραμμάτων τα οποία ε, ε, δημιούργησαν πρόβλημα όσον αφορά την συγχρηματοδότηση. Δηλαδή εμείς είδαμε ότι επιτόπου αντιμετωπίσαμε δύο ανταγωνιστικές καταστάσεις. Από τη μία τα εθνικά χρήματα και από την άλλη τα κοινοτικά χρήματα και βλέπετε σε, στο επίπεδο των περιφερειών ε, και των ε, δήμων μερικές φορές είναι δύσκολο ε, να διαχειριστεί κανείς μια κατάσταση όπου υπάρχουν δύο χρηματοδοτήσεις σημαντικές και επίσης θα πρέπει εκεί να γίνει κάποιος υπολογισμός για το ποια χρήματα μπορούν να είναι άμεσα διαθέσιμα, ποια είναι τα χρήματα τα οποία μπορούν και αργότερα να χρησιμοποιηθούν κτλ σε ορισμένες χώρες ε, είδαμε λοιπόν ε, κάποιο δισταγμό επιτόπου ε, για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Δηλαδή στην ουσία έλεγαν δεν μπορούμε να περιμένουν λίγο τα διορθωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουμε τα εθνικά χρήματα. Εν πάση περιπτώσει όμως πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία τελικά απεδείχθησαν ελάσσονος σημασίας νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι το τελικό συνολικό αποτέλεσμα έτσι όπως αντικατοπτρίζεται σε τις δαπάνες του επόμενου χρόνου, η εικόνα λέω είναι ε, καλή. Ε, και η τελευταία σκέψη την οποία θα ήθελα να κάνω αφορά το μέλλον. Το 2010 στην ουσία όλα τα εθνικά αντικυκλικά προγράμματα ολοκληρώνονται. Αυτό σημαίνει ότι από το 2011 και μετά δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα υπάρχει πολύ εθνικό χρήμα διαθέσιμο ε, για, ε, μεγάλες, για να καλυφθούν τα μεγάλα ελλείμματα. Και είναι σημαντικό ε, και είναι σημαντικό να προβλέψουμε λοιπόν ε, σε αυτήν, ε, αυτή την κατάσταση έτσι ώστε τα διαρθρωτικά ευρωπαϊκά ταμεία να διασφαλίσουν μια κατάσταση όπου ένας ελάχιστος βαθμός επενδύσεων θα εξακολουθήσει να υπάρξει. Και αυτό είναι δικό μας θέμα και το δουλεύουμε ήδη από φέτος. Να εξασφαλίσουμε ότι του χρόνου θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκταμίευση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που δίδονται επιτοπίως μέσω των διαρθωτικών πόρων και ότι με τον τρόπο αυτό μετά από ένα πρώτο γύρο συζητήσεων με τα κράτη-μέλη και με τους συναδέλφους μας στις διοικητικές και ε, εθνικές αρχές πιστεύουμε ότι ναι μπορούμε, ναι μπορούμε να φτάσουμε το στόχο αυτό. Και αν σας φέρουμε τώρα υπεραισιόδοξος, ίσως έχει κανείς στην αρχή του χρόνου το δικαίωμα να είναι υπεραισιόδοξος, Πιστεύω ότι το 2011 θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και πάλι τις δαπάνες μας κατά 25 έως 30%. Αν το επιτύχουμε τώρα αυτό, θα έχουμε πραγματικά ένα σημαντικό αντίκτυπο με την εργασία μας και κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρώπης για να μπορέσουν να στήσουν τα σχέδιά τους, ιδίως τα μεγάλα σχέδιά τους και πρέπει να σας πω και πάλι, επί τη βάση των τελευταίων πληροφοριών που έχουμε αποκομίσει, εγώ τίνω να είμαι αισιοδοξότερο σήμερα από ότι θα ήμουν πριν από τέσσερις ή πέντε μήνες. Βλέπω λοιπόν ότι όλες αυτές οι επενδύσεις που κάνουμε στην αρχή της χρονικής αυτής περίοδου, είτε σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των επενδυτικών σχεδίων, είτε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση συστημάτων ελεκτικών τα οποία λειτουργούν από την πρώτη στιγμή Αν συγκρίνω λοιπόν με αυτά που έχουν γίνει στους τελευταίους μήνες, αρχίζουμε πλέον να συλλέγουμε τη σοδιά των προσπαθειών μας. Η ιδέα μας λοιπόν θα ήταν να επανέλθουμε του χρόνου με μια ακόμα πιο ισχυρή χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό και μιλάω για το 2011, να συνεχίσουμε να αυξάνουμε <clears throat> αυτά τα ποσά το 2012 και εν καιρό να φτάσουμε μια κορύφωση το 2013. Και μετά από το 2013 θα αρχίσει να κατέρχεται η χρηματοδότησή μας. Εάν το επιτύχουμε λοιπόν αυτό θα έχουμε πράγματι επιτύχει να θεσπίσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά την προώθηση της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο άτομο, κύριε Πρόεδρε, προσωπικά. Επειδή είχαμε αυτή την ευκαιρία να καταδείξουμε ότι παρά το γεγονό ότι η πολιτική συνοχής είναι μια μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη διαρθρωτική πολιτική και αυτό το χαρακτήρα θα πρέπει να διατηρήσει. Παρ' όλα αυτά, κατέστη δυνατό μέσω μια κοινή προσπάθεια από την πλευρά και των περιφερειών των κρατών μελών καθώ και τη Κομισιόν να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέσα στη διαρθρωτική αυτή πολιτική για να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα περιφερειακής πολιτικής μέσα στα χρόνια της κρίσης. Επομένως, οι συνολικές μας πληρωμές το 2009 26,7 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και Συνοχή 25,4 δισεκατομμύρια και εξ αυτών 18,4 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2007-2013 και από αυτά τα 18,4 9 δισεκατομμύρια 9,4 δισεκατομμύρια μάλιστα 9 είναι προκαταβολές 1,4 ενδιάμεσες πληρωμές και μεταφερόμενα 6,2 δισεκατομμύρια τα οποία σιγά σιγά ε, αποπληρώνουμε στην αρχή του τρέχοντος έτους με μια αύξηση των δαπανών που προβλέπεται το 2010 και το 2011. Με τις αυξήσεις αυτές θα έχουμε πιο εποφελή αποτελέσματα για την οικονομική ανάπτυξη και θα είναι απαραίτητη αυτή η αύξηση για να συνεχίσουμε να δαπανούμε τον προϋπολογισμό με ένα αηφόρο ρυθμό και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά μου σχόλια. Θέλησα να σας περιγράψω το γενικό πλαίσιο και πάλι κύριε Πρόεδρε μεγάλη ευκαιρία για μένα να αναφερθώ στην Επιτροπή σας και είμαι έτοιμος να σας στείλω και ένα έγγραφο πληροφοριακό για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Σταυρακάκης. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά για την τόσο ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας. Αρχίζει τώρα η συζήτηση. Έχει το λόγο τώρα η κυρία Κρέελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Άνερ. Είναι πραγματικά κάτι που μας δίνει αισιοδοξία αυτό το οποίο λέτε, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός χρόνου, ο οποίος δεν είναι και τόσο φωτεινός. Εγώ θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση και την κατασκευή στεγαστικών καταλημάτων. Στα παλιά κράτη-μέλη υπήρχε ένας χαμηλός ρυθμός ε, χρησιμοποίησης αυτών των ε, ποσών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο λοιπόν εκταμιεύθηκαν αυτά τα ποσά, ιδίω στα παλιά κράτη-μέλη, θα ήταν σε μια εποχή οικονομικής κρίσης ένα πολύ καλό σχέδιο για τους Δήμους και τις κοινότητες να χρησιμοποιηθούν αυτά τα σχέδια, αλλά από ό,τι ξέρω στην περίπτωση της ε, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας ούτε ένα από τα ομόσπονδα κράτη έχει τροποποιήσει τα σχέδιά του για το τρέχον έτος, για το 2010. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η κατάσταση σε χώρες όπως η Γερμανία, στα παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, έχουμε περίπου 15 δισεκατομμύρια για τα 7 χρόνια τα επόμενα, τα τρέχοντα μάλλον, για την πολιτική συνοχής. Ε, 50 μάλλον εκατομμύρια τα 7 χρόνια, αλλά μου λέτε ότι 26 εκατομμύρια θα δοθούν το 2009. Κάπου δεν βγάζουν νόημα αυτοί οι αριθμοί για μένα. Δεν μπορώ να τα υπολογίσω σωστά. Πώς γίνεται αυτό. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Άνερ. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τον τομέα στέγασης, Πρόκειται κυρίως για πρόθεση κατοικιών που είναι ενεργειακά αποδοτικές. Είναι πολύ περιορισμένη η απορρόφηση των κονδυλίων προς το παρόν. Δεν έχουμε φτάσει λοιπόν αυτό το όριο του 4% το οποίο είχε θεσπιστεί. Βλέπουμε να υπάρχει ενδιαφέρον σε τα καινούργια αλλά και σε μερικά από τα κρατη όπως είναι η Γαλλία. και μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στα εθνικά προγράμματα. Κάποια κράτη-μέλη, κάποιες περιφέρειες εργάζονται τώρα για να προχωρήσουν να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους, τουλάχιστον αυτό αναμένουμε. Δεν νομίζω όμως ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε στο κατόφλι αυτό του 4% το οποίο προανέφερα. Και επειδή υπάρχουν αιτήσει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, να δούμε πότε θα το φτάσουμε αυτό το ποσοστό. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τη δική μας μεριά μια έρευνα στα κράτη-μέλη για να δούμε πότε φτάνεται αυτό το ποσοστό και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμο όλα αυτά τα μέτρα δεν έχει επιτευχθεί το ποσοστό του 4%. Πέραν όμως των μέτρων στα νέα κράτη-μέλη, πέραν του ενδιαφέροντος, <clears throat> πέραν των προθέσεων που εκδηλώνονται προς την κατεύθυνση αυτή από ορισμένα <clears throat> παλαιά κράτη-μέλη. Στην πράξη δεν υπήρξε μεγάλη αλλαγή. Τα 350 δισεκατομμύρια. Τα 26,7 τώρα που σας είπα ήταν τα χρήματα για την ε, πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική. Γιατί τα 350 δισεκατομμύρια μέσα στα 7 χρόνια περιλαμβάνουν και το κοινωνικό ταμείο μεταξύ άλλων. Αλλά στην πράξη έχουμε αργήσει ένα ολόκληρο χρόνο. Είμαστε περίπου στο 30% που έχουμε εκταμιεύσει για τη νέα αυτή περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι πολύ λίγα αυτά τα λεφτά Ακόμα και για λόγους λοιπόν προϋπολογισμούς είναι λίγα αυτά τα λεφτά, αλλά ακόμα περισσότερο για οικονομικούς λόγους είναι πολύ σημαντικό το να προωθήσουμε την εκταμείευση αυτών των ποσών και να συνεχίσει η πορεία. Είναι σαν την εκκίνηση ενός 747 που προχωράει πολύ αργά, σηκώνεται με μεγάλη δυσκολία και μετά πετάει πάρα πολύ ευχάριστα. Ελπίζω λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και στη συνέχεια. Αυτό το οποίο με ενοχλεί και αυτό το τονίζω πάντα όταν μιλάμε με τα κράτη-μέλη είναι ότι πράγματι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να απορροφηθούν τα κονδύλια μας από τις περιφέρειες, όχι από τα κράτη-μέλη αλλά θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά και μαζί σας για το τι θα κάνουμε σε σχέση με το, πρόβλημα της προσθετικότητας. Πολλά κράτη έχουν πολύ λίγα εθνικά χρήματα τα οποία μπορούν να, να κινητοποιήσουν από τον προϋπολογισμό τους Καλά κάνουν, τα χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για τον κοινό στόχο της πολιτικής συνοχής. Αλλά τι μένει τότε για να κάνουν αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν πρόσθετα. Πολλές χώρες λοιπόν αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης και αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει, ένα πρόβλημα που δεν έχει πάρει αοξία μορφή ακόμα, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε καλύτερα και να προετοιμαστούμε γιατί μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο προς το τέλος της περίοδου προγραμματισμού όταν θα δούμε πόσο καλά τηρήθηκε το κριτήριο της προσθετικότητας. Έχουμε καλούς λόγους λοιπόν σε επίπεδο προϋπολογισμού να συνεχίσουμε, αλλά έχουμε και οικονομικά επιχειρήματα τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να προβούμε σε αυτές τις επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ για, την... για τις πληροφορίες του κ. Γκουτμάν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο μόνιμος εισηγητής για το Ταμείο Συνοχής και είμαι σίγουρος ότι τα ίδια ερωτήματα που σας στέλνει η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα σας στείλει και η Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων. Τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα λαμπρά. Τρία ερωτήματα θα σας δώσω. Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε σήμερα, μπορείτε να μας δώσετε έγγραφη απάντηση. Πρώτον, είπατε από το 2002 ως το 2006 υπήρχε μια περίοδος προγραμματισμού η οποία παρατάθηκε για το Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. Η καταληκτική προθεσμία για να δοθούν τα δικαιολογητικά για τις ε, πληρωμές. Υπήρξε μια παράταση λοιπόν, αλλά αν δω τι έγινε με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία της 1ης Ιανουαρίου δείχνουν ότι 1,9 των χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε κάπου 4,2 δισεκατομμύρια. Γιατί αν τα κράτη-μέλη δεν έχουν δικαιολογητικά ως το τέλος Ιουνίου, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα απόδοσης <clears throat> των κονδυλίων αυτών. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Αυτά τα χρήματα μπήκαν στον προπολογισμό, δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν μπορούν να μεταφερθούν στα άλλα ταμεία και το ερώτημα είναι υπαριθμόν ένα. Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά. Ρώτησα και τον ε, υποψήφιο επίτροπο, τον κύριο Λεβεντόφσκι, για τα θέματα αυτά. Γιατί τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταμείο αλληλεγγύης, υπάρχουν άλλες δυνατότητε για τη χρησιμοποίησή τους. Ποια θα είναι η τύχη αυτών των χρημάτων. Γιατί βλέπουμε μια κατάσταση η οποία απολύτως δεν είναι καλύτερη. Και θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε. Τον Ιανουάριο του 2010 όλα τα ταμεία, η εκταμείευση λαμβάνοντας υπόψη και τις προκαταβολές και τις ενδιάμεσες πληρωμές για όλες τις χώρες ήμασταν στο 31%. Για 44% των κρατών μελών το ποσοστό είναι ακόμα χαμηλότερο. Και μερικά κράτη είναι 300% πιο χαμηλά από τα καλά κράτη. Αν δείτε το Περιφερειακό Ταμείο μπορούμε να δούμε Βλέπουμε η διαφορά μεταξύ των καλών και των κακών κρατών να είναι τέσσερις φορές, τέσσερα, επί τέσσερα. Αν δούμε το κοινωνικό ταμείο περαιτέρω, η διαφορά μεταξύ των καλών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και των καλών είναι απίστευτη. 469% πέντε φορές δηλαδή. Και είπατε το πρόβλημα είναι η ανάγκη χρηματοδότηση, ότι είναι ένα πρόβλημα προϋπολογισμού. Αλλά αν αναδυφίσει κανείς τον κατάλογο των χωρών που δεν έχουν ε, ικανοποιήσει τα κριτήρια είναι χώρες που δεν έχουν ελλείμματα, δεν έχουν προβλήματα στον προπολογισμό. Άλλοι λόγοι συνηγορούν λοιπόν για τη μη εκπλήρωση των κριτηρίων και τη μη εκταμίευση. Θα πρέπει λοιπόν να τροποποιήσουμε τα μέτρα μας γιατί αλλιώς θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση ως το 2002-2006 όταν προβλέπονται από τις προοπτικές αλλά τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται και πρέπει να ξαναγυρίσουν στα κράτη-μέλη και να μην χρησιμοποιηθούν για αυτό το στόχο. Γιατί εδώ αυτό είναι κακό, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα το οποίο δίνει προχρηματοδότηση, προκαταβολές κτλ. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε τώρα και τα δώσαμε σε άλλες γραμμές του προπολογισμού. Δεν είναι λοιπόν τόσο συστηματική αυτή η χρήση των χρημάτων. Τέλος για το 2010. Και αυτό είναι περισσότερο θέμα ελέγχου του προϋπολογισμού. Είπατε ότι έχετε επιτύχει καλή, καλό επίπεδο πληρωμών. Οι ενδιάμεσες πληρωμές όμως δείχνουν ότι σε 27 ημέρες από την 1η Νοεμβρίου ως την 1η Δεκεμβρίου αυξήσατε κατά 37% το κοινωνικό ταμείο και 55% για το ταμείο το περιφερειακό και το ταμείο συνοχής. Όλα αυτά τα πλήρωσε η Κομισιόν σε 27 μέρες. Είτε έχετε μαζέψει τα δικαιολογητικά από τα κρατημένη και περιμένατε να τα πάρετε όλα, τα αναλύσατε και μετά πληρώσατε, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αλλά αν τα κρατημένη μαζέψαν όλα, όλα αυτά τα χαρτιά και σας τα φέραν στο κεφάλι και σας είπαν πληρώστε τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου και έπρεπε να τα πληρώσετε για να μην επιτύχετε, για να μην πέσετε σε ρυθμό εκταμίευσης, αυτό θέτει πολύ σοβαρά ερωτήματα ποιότητος σε σχέση με το λογιστικό έλεγχο και σε σχέση με την δημοσιονομική πειθαρχία. Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε σήμερα, απαντήστε αύριο ή μεθαύριο ή εγγράφος. Αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η πληροφορία. Αυτά πρέπει να μας τα δώσει η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Καταρχήν, επιτρέψατε μου να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας δώσω άμεσα μία απάντηση. Οι χώρες μέλη πράγματι πληρώνουν τους λογαριασμούς που λαμβάνουν, κάνουν τους αναγκαίους ελέγχους και πληρώνουν τους λογαριασμούς που λαμβάνουν στο επίπεδο των διαχειριστικών αρχών. Στη συνέχεια συγκεντρώνουν όλες αυτές τις ε, απαιτήσει, τις ε, επανεξετάζουν και μέσω των ε, οργάνων που διαθέτουν και αυτή τη στιγμή γίνει αυτή η πιστοποίηση. Μας αποστέλουν έναν αριθμό των πληρωμών που έχουν συγκεντρώσει που στη συνέχεια επανεξετάζονται στην περίπτωσή μας και στις 27, στο διάστημα των 27 ημερών που αναφέρατε έχουμε καθαρίσει όλους αυτούς τους, όλες αυτές τις πληρωμές και υπάρχει ένας πρώτος ταχύς έλεγχος και εάν δεν έχουμε διαπιστώσει πρόβλημα. Εκείνες οι πληρωμές όπου ανακύπτουν κάποια προβλήματα ή πρέπει να διευκρινιστεί ένα επιπρόσθετο θέμα μεταφέρονται στο 2010, δεν αποπληρώνει το 2009 και οι περιπτώσεις αυτές διευκρινίζονται με τις χώρες μέλη ούτε ώστε να εξασφαλίσουμε όταν, ότι όταν αποπληρώνουμε, επιστρέφουμε τα ποσά αυτά, αυτό γίνεται ε, έχοντας την αίσθηση, την εξασφάλιση ότι τα πράγματα είναι εντάξει. Αλλιώς ε, διενεργούμε τους συνήθεις έλεγχους ελέγχους από τα εποπτικά όργανα, από τα ελεγκτικά όργανα. Όπως σας είπα, όταν έχουμε κάποια ποστά εκπλήρωση της τάξης του 30% κατά μέσο όρο, ε, εγώ δεν είμαι σύντος, ε, περήφανος γι' αυτό, γιατί υπάρχει καθυστέρηση ενός ε, έτους στην περίπτωση αυτού, αυτή. Και αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα πρέπει να καταβάλουμε όλες τις αναγκαίες προσπάθειες από τη δική μας πλευρά για να καλυφθεί αυτή η καθυστέρηση. Και ένα τμήμα αυτών των προσπαθειών είναι ότι εμείς από την πλευρά μας θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και θα βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή με εκείνες τις χώρες μέλη και περιφέρειες όπου τα ποσοστά εκπλήρωση είναι ιδιαίτερως χαμηλά, όπως αναφέρατε. Και υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, αρκετές περιπτώσεις, όπου ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτές τις επαφές, γιατί κατά τη διάρκεια του 2009 διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν με ένα βραδύτερο ρυθμό. Και καμιά φορά ε, πρόκειται για θεσμικούς ε, λόγους, για παράδειγμα, και κυβερνήσεων, ε, οφείλονται στην τύχη, αλλαγέ κυβερνήσεων, νέοι αξιωματούχοι, νέοι υπουργοί, νέοι γενικοί γραμματεί αναλαμβάνουν καθήκοντα και έτσι σημειώνονται τι τις Αλλά καμιά φορά υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αυτά πρέπει να εξετάσουμε κατά περίπτωση γιατί τα ποσοστά εκπλήρωση είναι τόσο χαμηλά και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το ποσοστό αυτό να αυξηθεί ακόμα και σε εκείνες τις χώρες που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση που βρίσκονται πίσω. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό γύρει και άλλα ερωτήματα, δεχομένω πολιτικά ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να θέσουμε επιτάπητος. Τώρα, όσον αφορά το 1,9 της, της περιοδου 2000-2009, τα χρήματα αυτά έχουν διασωθεί. Για το 2000-2006 η Επιτροπή ε, μπορεί να πληρώσει μέχρι το 95%. Υπάρχει μια οροφή λοιπόν την οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει η Επιτροπή. Είναι το 95%. Με πρακτικούς όρους για όλα τα προγράμματα που έχουν πετύχει το 95% το ποσό αυτό έχει παγώσει μέχρι να λάβουμε όλα τα έγγραφα. Τα ποστά αυτά θα αποδεσμευθούν. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίε τη Επιτροπή έχουν αναλύσει την οριστική έκθεση εφαρμογή, την ε, δήλωση που έχει, και που έχει παράσχει το ε, όργανο ελέγχου, το ελεγκτικό όργανο. Ε, τα ποσά αυτά θα εκτελεστούν μόνο εφόσον λάβουμε τα τρία έγγραφα και αυτή τη στιγμή η Επιτροπή τα έχει αναλύσει και έχει διαπιστώσει την ορθότητα, ξεκριβώς την ε, ορθότητα των αριθμών, των στοιχείων. Τα ποσά αυτά θα πληρωθούν μόνο αυτή τη στιγμή λάβουμε αυτά τα έγγραφα. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω ότι έχουμε λάβει ορισμένα έγγραφα από τις χώρες μέλη And this amount was released for Και αυτά τα ποσά θα αποδεσμευθούν, θα κατανοηθούν για αυτές τις χώρες. Είναι φυσιολογικό λοιπόν, υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ναι, εγώ δεν μιλάω για 95% ποσοστό εκπλήρωσης που θα πληρωθούν από την Επιτροπή όταν κλείσουν τα έγγραφα. να δούμε τα αποστά εκπλήρωση για το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης την 1η Ιανουαρίου αυτού του έτους μπορείτε να δείτε μισό χρόνο μετά την εκνοή της προθεσμίας η ιανουαριου αυτου του ετου μπορειτε να δειτε μισο χρονο μετα την εκνοη τη προθεσμιας η εκπληρωση δεν ανέχει στο 95%, στο 92%, στο 93% και η διαφορά μεταξύ των 95% και των 92% είναι 3% δεν μπορώ να δω πώς θα μπορεί να εκπληρωθεί το 3%. Γιατί αν δεν είμαστε έτοιμοι να παράσουμε τα έγγραφα αυτά τον Ιούνιο του περασμένου έτους, τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να σωθούν τόσο εύκολα. Δεν μιλάω για το 95% όπως τα εκπλήρωσε εδώ, η περίπτωση είναι ξεκάθαρη. Το ποσοστό ήταν 60 δις τέλος του προηγούμενου έτους και είναι σαφές ότι τα 5% θα πληρωθούν από αυτά τα δίσε αλλά για εκείνα τα μια που έχουν κλείσει υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί γιατί τα ποστά εκπλήρωση δεν ήταν 55% μετά την εκμονή της προθεσμίας και αυτό είναι το ερώτημα που έθεσα Ωραία, επιτρέψατε μου να διευκρινίσω αυτή την κατάσταση. Ε, το 95% η περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρη. Λοιπόν, πληρώνουμε μέχρι το 5% και κρατάμε 5% για το κλείσιμο και αυτή τη στιγμή έχει γίνει το κλείσιμο. Αυτά τα 5% αποδεσμεύονται. Εάν απομείνουν κάποια χρήματα οποία δεν έχουν πληρωθεί, δαπανηθεί, τα χρήματα αυτά έχουν σωθεί. Τα χρήματα αυτά, συνεπώς, δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλα προγράμματα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν από την άλλη εν υπάρχουν επενδυτικά προγράμματα τα οποία υπερβαίνουν μια περίοδο των 7 ετών, νομίζω ότι αναπόφευκτα θα φτάσετε σε ένα σημείο που υπάρχουν πάντοτε προγράμματα τα οποία δεν λειτουργούν. Προγράμματα που δεν λειτουργούν, όπως είπα, και αν φτάσουμε σε ένα εσφαλμένο 99% στο τέλος, εγώ προσωπικά δεν το έβρισκα και τόσο κακό. Αλλά βεβαίως ε, θα σας δώσουμε μια απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα που θέσατε. Και πάλι θα ήθελα να πω ότι έχετε δίκιο. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι την επόμενη περίοδο, το 2007-2013, τα χρήματα να δαπανώνται τόσο καλά όσο είναι δυνατόν, όσο μπορούμε να πετύχουμε δηλαδή. Και τώρα βρισκόμαστε στην αρχή της περίοδου όπου ανακαλύπτουμε μια σειρά προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι σαφές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σρέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις κυρία Άνερ. Καταρχήν καλώς ήρθατε εδώ και θεωρώ σημαντικό να μας δίνετε αναφορά για την διαδικασία που θα αντικοποιήσουμε προσεχώς. Έχω μία ερώτηση σε σχέση με τα όσα παρουσιάσατε, η οποία πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση, όπως ε, χάραξε ο σας. Εάν ε, μιλάμε για τόσο μεγάλα ποσά πώς διενεργείται ο έλεγχος ποιότητας. Μας είναι ιδιαίτερος σημαντικό να τηρείτε το δίκαιο του περιβάλλοντος, να πρόκειται για βιώσιμες επενδύσεις, πραγματικά εξυπηρετούν τα συμφέροντα των περιφερειών και όχι όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από πέντε χρόνια να κλείσει επιχείρηση, να φύγει από εκεί κλπ. Ε, γιατί ναι μεν έχει γίνει μια προετοιμασία σε μια περιοχή αλλά τελικά ε, δεν εμφανίζεται κανείς και λοιπά. Κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ε, ποια, ποιους άμεσους ελέγχους έχετε στη διάθεσή σας ούτως ώστε να εμποδίσετε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν ένα πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια της βεσιμότητας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το μέλλον. Χθες ε, ε, μας είπε η Ισπανική Προεδρία ότι συνήλθε μια επιπρόσθετη ομάδα υψηλού επίπεδου της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα εν σχέση με το τι έγινε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Άνερ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν το θέμα της, ε, του ελέγχου ποιότητας ε, για τα ποσά αυτά. Υπάρχουν τρεις ε, τύποι ελέγχου που είναι άμεση και υπάρχουν και κάποια άλλοι έλεγχοι που γίνονται πιο μακροπρόθεσμα. Άμεσα υπάρχει μια υποχρέωση για τις διαχειριστικές αρχές στο σύστημα της κοινή διαχείρισης που έχουμε ε, κάνουμε μια διάκριση δύο τύπ, μεταξύ δύο τύπων προϊόντων. Ε, δύο τύπων προγραμμάτων. Τα συνήθι προγράμματα, τα οποία είναι κάτω από 25 ή 50 εκατομμύρια ευρώ και τα μεγαλύτερα, τα μεγάλα προγράμματα. Όσον αφορά αυτά τα μεγάλα προγράμματα, όταν πρέπει να παρουσιαστούν στην Επιτροπή, εξετάζονται από τις περισσίες της Επιτροπής όσον αφορά και το βαθμό συμμόρφωσης με την κοινωτική νομοθεσία, με όρους περιβάλλοντος, ε, τις δημόσιες προμήθειες κλπ. Τα άλλα προγράμματα επιλέγονται ε, ε, στη βάση της ευθύνης των αρχών αυτών διαχείρισης μαζί με τις επιτροπές παρακολούθησης της χώρες μέλη και στις περιφέρειες. Και εδώ έχουμε καταρχήν τους ελέγχους που ενεργούν οι διαχειριστικές αρχές για αυτά τα προγράμματα. Το όργανο πιστοποίησης πριν αποστείλει τις αποτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει κάποιους ελέγχους για να εξακριβώσει κατά πόσα έκαναν σωστά διαχειριστικές αρχές το έργο τους και θα υπάρχουν και ετήσιες εκθέσεις οικονομικού ελέγχου από τις χώρες μέλη που πρέπει να ελέγξουν, οφείλουν να ελέγξουν τα διάφορα προγράμματα. Αυτό είναι που συνήθως έχουμε, κάνουμε όταν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για τις πληρωμές. Και αφού ε, κάνουμε και εμείς μια σειρά οικονομικών ελέγχων ε, και το ελεγκτικό συνέδριο από την πλευρά του εξετάζουμε το βαθμό συμμόρφωσης. Αυτό το οποίο δεν εξετάζομαι στη φάση αυτή είναι ε, ποια είναι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Και αυτό μου κάνει τη γέφυρα με, την, με το θέμα θίξατε για την ομάδα υψηλού επίπεδου και χθεσινή συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει θα σας δώσουμε μια πιο λεπτομεριακή ε, παρουσίαση. Η Κατερίνα Μαρτινόβα που είναι πρόεδρος της ομάδας της θα σας μιλήσει. Χθε η συνεδρίαση αυτή είχε απαιτείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα έγιναν κάποιες γενικότερες συζητήσεις σχετικά με την, Ευρώ, με την Ατζέντα Ευρώπη 2020 που παρουσίασε ο πρόεδρος ε, Μπαρόζο και ε, παρουσιάστηκε προς τους συναδέλφους των χωρών μελών και η συζήτηση είχε σαν σκοπό να δείξει σε ποιο βαθμό μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το μελλοντικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ευθυγραμμίζεται με αυτό το στόχο. Ποιο είναι το περιθώριο ευελιξίας που χρειαζόμαστε για να αφήσουμε στις περιφέρειες και στις ενδιαφερόμενες χώρες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν όχι μόνο στους κοινού στόχους, αλλά επίσης και στις, στα, ειδικά, τοπικά, στα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα. Το θέμα της ευελιξίας λοιπόν ε, συζητήθηκε, έπαιξε μια ανταλλαγή απόψεων, δεν ε, υπήρξαν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και επίσης χθε είχαμε την ε, παρουσίαση των συναδέλφων από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Γενική Διεύθυνση Γεωργίας που παρουσίασαν τα δικά τους οράματα για την μελλοντική ανάπτυξη των δικών τους ε, πολιτικών πεδίων που πιστεύω συνδέονται στενά με την ε, δική μας πολιτική, την περιφερειακή πολιτική δηλαδή. Και εδώ είχαμε κάπως πιο γενικές παρουσιάσεις και εδώ θα πρέπει σίγουρα να δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες με τους συναδέλφους πώς μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση γιατί έχουν ακριβώς κατά νου. Χθε το απόγευμα έγινε μια συζήτηση, είχα μια συζήτηση με τους συναδέλφους των χωρών μελών σε σχέση με το πώς μπορούμε να εισαγάγουμε μια καλύτερη αξιολόγηση της ποδοτικότητας της πολιτικής μας κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όχι δηλαδή εκ των υστέρων αξιολογής, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι μια επιχείρηση ε, πραγματικά ανταποκρίνεται στην ποιότητα των προγραμμάτων ή τι αποδίδουν τα προγράμματα αυτά όσον αφορά την περιβαλλοντική ε, προστασία, όσον αφορά την ανταπόκριση στο περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα όπου είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων χθες και ασφαλώς αυτό θα συνεχίσει να μας απασχολεί στο πλαίσιο της συζήτησης σχέση με τους μηχανισμούς της δικής μας ε, πολιτικής συνοχής. Πώς μπορούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται επί τόπου και ιδιαίτερως εκείνα τα προγράμματα για τα οποία δεν έχουμε άμεση γνώση, δηλαδή όχι τα μεγάλα προγράμματα, αλλά τα υπόλοιπα. Κατά πόσο είναι ικανοποιητικό αυτό το οποίο γίνεται επί τόπου για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Αυτό είναι ένα σημείο όπου θα πρέπει να συζητήσουμε κάποιες ιδέες που ανέκυψαν και από την ίδια τη συζήτηση. Και θα ήθελα να συζητηθώ με τους συναδέλφους. Αν μου επιτρέπετε, θα επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί ήδη κάνατε μια συνεδρίαση για την αξιολόγηση. Και νομίζω το πραγματικό ερώτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το πώς κατά τη διάρκεια ενός περίοδου μπορούμε να εξασφαλίζουμε την ποιότητα μέχρι στιγμής κάνω μια εκ των υστέρων αξιολόγηση, αλλά θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα βεβαίω από αυτό, αλλά κυρίως να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, κατά τη διάρκεια της περίοδου που τρέχει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο <clears throat> κύριος Όλμπρεχτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις έχω και δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, για το ερώτημα που έθεσε η Κωνσταντ Κρέελ. Είναι σαφέ για οποιονδήποτε ο οποίος γνωρίζει τις περιοχές αυτές ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη γνώση για τα θέματα αυτά της ε, αποδοτικότητας για την ενέργεια. Αν αλλάζουμε συνέχεια τους κανόνες κατά τη διάρκεια της περίοδου προγραμματισμού και στην αρχή δίνουμε σαφείς κανόνε, αλλά λέμε στη μέση του δρόμου ότι μπορείτε να αλλάξετε του κανόνε. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το λειτουργικό πρόγραμμα, γιατί κάπου θέλουν να πάρουν τα χρήματα. Και επομένως φτάνουμε στο τέλος της χρονικής περίοδου και τα χρήματα δεν δαπανώνται. Οπότε ακόμα και ο πιο σημαντικός στόχος για το περιβάλλον που είναι η ενεργειακή απόδοση των σπιτιών δεν θα υλοποιηθεί. Το ερώτημα είναι, είμαστε έτοιμοι να βρούμε νέα λεφτά για να προωθήσουμε τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια. το να αλλάξουμε πολιτικά το λειτουργικό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουμε από την πράξη, γιατί ρωτούμε όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται επί το τους λέμε από πού να πάρουμε τα λεφτά. Και τώρα τι θα γίνει με τα λειτουργικά προγράμματα στο μέλλον. Ίσως μπορούμε να κάνουμε πιο ανοιχτό, πιο ευέλικτο το σύστημα αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να μα πει το ελεκτικό συνέδριο ότι όλα αυτά δεν είναι ελέγξιμα. Μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, όπως και η διαμοιρασμένη διαχείριση. Τα κράτη-μέλη δεν δαπανούν τα χρήματα και τώρα λένε γιατί η Κομισιό δεν κάνει κάτι να δαπανίσουν τα κράτη-μέλη τα χρήματα. Ίσως η Κομισιό πρέπει να ξανασκεφτεί το ρόλο το οποίο διαδραματίζει. είναι απλώ εποπτική η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φταίνουν τα κράτη-μέλη ή πρέπει να είναι πιο παρούσα επιπλέον η Επιτροπή. Γιατί είτε το βλέπουμε αυτό σαν επενδύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δαπανά τα χρήματα, ή εναπόκειται στα κράτη-μέλη τα οποία δεν δαπανούν τα χρήματα και τότε δεν έχουμε τρόπο δράση. Πριν από πέντε χρόνια προσπαθούσαμε να προτείνουμε να αναχρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά τα οποία δεν θα ήταν εκταμιευμένα για την πολιτική συνοχής. Αλλά ούτε το Συμβούλιο ούτε η Κομισιόν δέχτηκαν να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τότε αν συγκρίνουμε με το παρελθόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1,5% είναι μια μεγάλη πτυχία. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε δυσκολίες με την Επιτροπή μας τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα ήταν χρήσιμο να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για να μας εξηγήσετε γιατί έχουμε αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε τους αριθμούς, αλλά θέλουμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δύο ερωτήσεις. Μία είναι πιο γενική. Η οικονομική κρίση έχει βοηθήσει την πολιτική συνοχή ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν τα δικά τους εργαλεία Όλοι ξέρουν λοιπόν ότι τώρα είναι δυνατό να γίνει αυτή η πολιτική όχι μονάχα με ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά με εθνικά χρήματα. Έχουμε λοιπόν μια νέα κατάσταση. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής θα επανααναλυθεί μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης για να βρεθούν οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι τυχαία, κάτι θα πρέπει να αλλάξει λόγω της μεθόδου που μπορεί να ακολουθηθεί από τα κράτη-μέλη τα λεγόμενα ευκολότερα χρήματα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος το ερώτημα, το τελευταίο μου ερώτημα έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Αν έχουμε προβλήματα σήμερα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά στους προϋπολογισμούς του 2011, 2012 και επέκεινα. Κάποιοι από εμά είναι και μέλη τη Επιτροπή Προπολογισμού. Η τάση μα είναι να μειώνουμε τα χρήματα στον προπολογισμό, γιατί αν δεν εκταμιεύονται, τότε τον επόμενο χρόνο βλέπουμε ότι δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά χρήματα. Ποια είναι λοιπόν η θέση της Γενικής Διεύθυνσης για τα περιφερειακά θέματα σε σχέση με τον προϋπολογισμό αν μειώνουμε τους προϋπολογισμούς, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια πολιτική συνοχή για να είναι πιο έντονη από ό,τι σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Άνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με την ε, πραγματική ερώτηση όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να δούμε τον προϋπολογισμό 10, 11, 12, 13. οι προβλέψεις μας ε, και τα, τα προγράμματά μας, τα οποία βεβαίως εξαρτώνται και από τις δραστηριότητες, είναι να έχουμε σταθερή αύξηση του προϋπολογισμού έτσι ώστε το 2013 να φτάσουμε στο ψηλότερο σημείο. Όμως αυτό θα πρέπει να οργανωθεί με τρόπο ώστε το 2013 όταν θα φτάσουμε στην κορυφή να μην έχουμε ξεπεράσει την οροφή ε, του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι καταβάλλονται ήδη από το 2010 και το 2011 όλες οι απαραίτητες προσπάθειες έτσι ώστε στα ε, προγράμματα τα οποία ε, λαμβάνουν χώρα επιτόπου να υπάρχει και η πρόβλεψη για τα επόμενα προγράμματα. Αυτή η program pipeline όπως ε, τη λέμε. Ήδη το δουλεύουμε το σύστημα αυτό και μιλάμε για μία αύξηση, αν μιλάμε δηλαδή 25-30% ε, θα έχουμε και αύξηση αντίστοιχη για το 2012 και το 2013 και μετά το 2013 θα έχουμε φτάσει στην κορυφή λοιπόν γιατί θα έχουμε το 1 συν 2, 1 συν 3 ε, ε, που θα ισχύει και για τις νέες χώρες και μετά το 2013 ενδεχομένως θα έχουμε μία ελαφρά καθοδική πορεία για για το σύνολο της ε, περίοδου ή θα δούμε πώς μπορέσουμε να μείνουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, το, σημείο, το σημαντικό είναι ότι, μέχρι, ότι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την διαρκή αύξηση θα πρέπει να έχουμε επενδύσεις επιτόπου και νομίζω ότι η εντύπωσή μου είναι τελικά ότι η κρίση ενδεχομένως θα έχει θετικό αποτέλεσμα για την πολιτική συνοχής. Όχι γιατί η πολιτική συνοχή μπορεί να θεωρηθεί πολιτική αντιμετώπιση κρίσης. Δεν είναι αληθές αυτό. Όμως πρόκειται για μία μακροπρόθεσμη ε, πολιτική και αυτό που καταδεικνύεται από τις συζητήσεις τώρα είναι ότι ενδεχομένως υπάρχουν ε, σε αυτή αυτή τη χρονική διάρκεια που μας ε, ενδιαφέρει, κάποια σημεία κρίσης, ε, αλλά ε, παρόλα αυτά μας δίνεται η δυνατότητα βάσει των των εργαλείων να τις αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις αυτές. Και ένα άλλο σημαντικό είναι ότι μετά το 2010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 να προχωρήσουν με ε, δαπάνες μέσω ελλείμματος θα μειωθεί ακόμα περισσότερο. Ε, πέραν αυτού βεβαίως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα και για πολλές χώρες ε, αυτά τα χρήματα θα αποτελέσουν μια βάση στήριξης και εν πάση περιπτώσει οι Υπουργοί Οικονομικών προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα χρήματα αυτά σαν αποθεματικό. Τους ενδιαφέρει γιατί αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο ε, για τις επενδύσεις. Και ένα άλλο σημαντικό πράγμα. Τη στιγμή που αυτές οι επενδύσεις ε, τις θέλουμε και θέλουμε να είναι προσανατολισμένες προς το μέλλον ε, και να είναι ευθυγραμμισμένες με τους δικούς μας στόχους δηλαδή της βελτίωσης ε, της ε, ανταγωνιστικότητας, προσαρμογής της κλιματικές αλλαγές, ε, προώθησης της πράσινης οικονομίας κλπ. <clears throat> Και βεβαίως αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα υπογραμμίσουμε τα επόμενα χρόνια και μάλιστα προτιθέμεθα να ε, κάνουμε δύο ανακοινώσεις ε, φέτος. Ε, η πρώτη θα αφορά την κοινωνική συνοχή και την εφορία και το δεύτερο θα αφορά την διασύνδεση ανάμεσα σε καινοτόμες επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή. Δύο ανακοινώσεις λοιπόν, οι οποίες θα μας εμπνέουν και για τις μελλοντικές μας δραστηριότητες. Βλέπουμε βλέπουμε ότι βαθμία όλο και περισσότερες χώρες, όλο και περισσότερες ε, περιφέρειες ε, προετοιμάζονται να αλλάξουν τα προγράμματα, τα προγράμματά τους. Πρέπει να σας πω ότι σε πολλές περιφέρειες πέρσι δεν τροποποιήθηκαν ε, τα προγράμματα γιατί θα χάνατε ακόμα έξι μήνες και το προτείναμε και εμείς, είπαμε εντάξει εφαρμόστε τα προγράμματα και θα δούμε μετά. Ε, αν μπορούν να γίνουν κάποιες τροποποίησεις. Τώρα όμως διαπιστώνω ότι έρχονται διάφορες επιστολές όπου οι ενδιαφερόμενοι μας ζητούν ε, σύμφωνη γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις προγράμματος. Ε, σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα και θα δούμε λοιπόν εάν αυτά τα επιδοτούμενα προγράμματα μπορούν να γίνουν αποδεκτά γιατί ακολουθούν την οδό της καινοτομία και της πράσινης οικονομίας. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε και προς τα κράτη και προς τις περιφέρειες. Το ξαναλέω λοιπόν αυτό, όμως θα ξαναπώ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν συγκεκριμένα προγράμματα σε συγκεκριμένες περιφέρειες τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και δεν μπορεί να έχουμε σωστή και ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη αν δεν αναπτύξουμε και τα προβλήματα, αν δεν αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα αυτά. Επομένως θα πρέπει να παραμείνει και ένας βαθμός ευελιξίας. Δεν μπορεί τα προγράμματα να είναι 100% για καινοτομία. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να παραμείνει και ένα ποσοστό ευελιξίας, αλλά βεβαίω αυτό θα το συζητήσετε και με το μελλοντικό επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσω τον λόγο στον κύριο Φανίστελ Ρόι. Έχω τέσσερις ομιλητές και έχουμε χρόνο μέχρι τις 10.30. Προσπαθήστε λοιπόν να είστε σχετικά σύντομοι. Ο Φανίστελ Ρόι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να εκπληρώσω την να τηρήσω μάλλον την ε, σύστασή σας. Έχω μία ερώτηση και μία πρόταση. Η ερώτηση αφορά την ανησυχία που έχει η Επιτροπή μας για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Μας πληροφόρησατε για τα στοιχεία, για τη γενική κατάσταση και συγχρόνως και θα συνεχίσει και η πορεία της διαδικασίας με την προετοιμασία της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Εμείς είδαμε ότι ήταν μια ψεύδο ενδιάμεση ή ενδιάμεση ψεύδο αναθεώρηση καλύτερα. γιατί υπήρξε μεταφορά χρημάτων από μια κατηγορία σε μια άλλη κατηγορία και έτσι λύνονται τα προβλήματα. Μπορείτε όμω να μα πληροφορήσετε για αυτή τη διαδικασία και για τον τρόπο με τον οποίο εσεί ω Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Θεμάτων εμπλέκεστε σε αυτή την υπόθεση. Είναι ένα πολιτικό θέμα. Μήπω θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πάρει την πρωτοβουλία να οργανώσει μια σημαντική ακρόαση για τη λειτουργία της πολιτικής συνοχής τα τελευταία χρόνια και αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την συνάντηση που έχουμε με τα Εθνικά Κοινοβουλία για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε μια συζήτηση μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και με αυτούς οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στα Εθνικά Κοινοβούλια για το μέλλον της πολιτικής συνοχής σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Μια πολύ επιπαιδική λοιπόν προσέγγιση μπορείτε να μας πληροφορήσετε λοιπόν για την εξελίξη διαδικασία και να μας κρατήσετε ενήμερους ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον και δεύτερον είσαστε έτοιμος να συνδυάσετε αυτέ τις διαδικασίες με κοινοβουλευτικές εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άνερ. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο που θέσατε μέσα στους κόλπους της Κομισιόν η συζήτηση είναι εν εκτιλήξη σε σχέση με το έγγραφο Ευρώπη 2020. Έγινε διαδικασία διαβούλευσης, υπήρξε ισχυρή συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης και προσωπικά χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας πω ότι η πιο σημαντική οντότητα η οποία συμμετέσχε σε αυτήν την διαδικασία ήταν οι περιφέρειες <clears throat> και οι περιφερειακές ενώσεις. Και οι συνάδελφοι από την Γενική Γραμματεία της Κομισιόν μας ζητήσαν να τους βοηθήσανε να τους βοηθήσουμε για να εξετάσουμε τα έγγραφα, τα έγγραφα διαβούλευσης τα οποία υπέβαλαν οι περιφέρειες και νομίζω ότι ήταν σαφής η θέση των περιφερειών. Καταρχήν υπογράμμιζαν το ρόλο των περιφερειών ως μοχλών ανάπτυξης, ως σημαντικών παικτών στην πολιτική αυτή <clears throat> και υπογράμμιζαν επίσης και τη σημασία της πολιτικής συνοχής <clears throat> σαν ενός θετικού τρόπου να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους που βρίσκονται στο έγγραφο Ευρώπη 2020. Η διαβούλευση αυτή <clears throat> είναι υπό εξέταση. Είναι πολλές άλλες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει από κράτη-μέλη, από επιχειρήσεις, από γενικότερα εμπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι, κράτη, ότι η Γενική Γραμματεία προσπαθεί να συντάξει μια σύνοψη και συγκέντρωση των απόψεων αυτών και ελπίζω ότι η νέα Κομισιόν όταν με το καλό αναλάβει τα καθήκοντά της θα δράσει ταχαίως. Αυτό θα σήμαινε ότι αρχές Μαρτίου <clears throat> θα μπορούμε να έχουμε αυτό το έγγραφο για την Ευρώπη 2020 που θα αποτελέσει και σημείο αναφοράς για το έργο μας σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της αναθεώρησης του προϋπολογισμού, περιμένω ακόμα να υπάρξει κάποιο έγγραφο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά Ίσως του χρόνου μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου πέρα των αναλογισμών για τον προϋπολογισμό και τις δημοσιονομικές προοπτικές θα χρειαστεί να φτάσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα αριθμητικά ποσά για το τι θέλουμε να κάνουμε στον τομέα της δράσης μας. και ο κύριος Χάν, που είναι ο μελλοντικό επίτροπος μάλλον, έχει τονίσει ότι έχει μια σαφή άποψη σε ό,τι αφορά τη συνολική αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής. Από τη δική μας πλευρά ακολουθούμε τις απόψεις του μαζί με τους συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού για το έργο που αφορά τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους για το θέμα της διακυβέρνησης και των συναφών πτυχών σε σχέση με, τους, με την Ευρώπη 2020. Και η θέση μας είναι πολύ σαφής. Είναι σαφές ότι σε τελική ανάλυση θα έχουμε μια πρόταση από το Σώμα των Επιτρόπων και ενδεχόμενες διαμεσολαβήσεις, arbitrage που θα πρέπει να γίνουν σε αυτό το επίπεδο. Και εν παραλίλω συνεχίζουμε το έργο με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες και με τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτήν την ε, υποδομή που βρίσκεται με το Γραφείο των Περιφερειών εδώ στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα με όλες τις ε, περιφέρειες και η πρότασή μου κύριε Πρόεδρε, αλλά πιστεύω ότι θα είναι και μια πρόταση η οποία θα ισχύει και για το μέλλον. Όταν έρθει και ο επερχόμενος επίτροπος να μιλήσει για το ε, πρόγραμμά του, είναι ότι θα ήταν πολύ θετικό να βρισκόμαστε σε συνεχή και στενή επαφή μαζί σας και μπορούμε να σκεφτούμε λοιπόν αν θα έπρεπε να έχουμε και μια μικρή ομάδα η οποία θα συνεργαστεί για τα θέματα αυτά. Μπορεί να σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό λοιπόν να το εξετάσετε μεταξύ σας. Εμείς από τη δική μας πλευρά είμαστε απόλυτα έτοιμοι να κάνουμε <clears throat> την παροχή τεχνικών πληροφοριών και να σας παρουσιάσουμε τις αναλύσεις οι οποίες είναι στα χέρια μας να τις κάνουμε διαθέσιμες σε εσά. Πρόβλημα δεν αποτελεί αυτό. Πιστεύω ότι με μεγάλη οκίτητα θα μπορέσουμε να φτάσουμε και στα πιο συγκεκριμένα στοιχεία του μέλλοντος Ζητώ λιγάκι την κατανόησή σας ως Γενικός Διευθυντής. Γιατί έχουμε βρεθεί σε μια κάπως δύσκολη κατάσταση του να να έχουμε μια σειρά από τρεις επιτρόπους, ο ένας έχει φύγει, ο ένας εργάζεται ακόμα και ο επόμενος θα έλθει από το Φεβρουάριο αλλά θα πρέπει πράγματι να μιλήσω με τον κύριο Χάν για να μπορέσει να αναπτύξει και αυτός τις απόψεις του για τη μελλοντική πολιτική γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο αρμόδιος επίτροπος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και είναι απόλυτα φυσιολογικό να είναι αυτός ο οποίος θα έχει να μας πει κάτι σε σχέση με το πώς θα πρέπει να Διαφανεί το μέλλον. πεπισμένο. είμαι βέβαια ότι θα χαρεί πάρα πολύ να έρθει ενώπιον σα και να συζητήσει με μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για τα θέματα αυτά και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε πιο συγκεκριμένα θέματα της πολιτικής αυτής που είναι τόσο σημαντικά όσο και η συνολική αρχιτεκτονική, τα συνολικά λοιπόν θέματα του πώς θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που θα είμαι στη διάθεσή σας για να συνηθίσω, μάλλον να συζητήσω τα θέματα αυτά μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία παρουσιάστηκε και υπογραμμίσατε. Ο ε, Στόιρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην μέση διάταξή μας υπάρχει και η έκθεση για το έτος 2009 και αυτό συνάπτεται με τα ερωτήματα που ανέφερε και ο κύριος Γκούτμαν. Είναι ένα ιδιαίτερο έτος το 2009 ή όλα αυτά είναι αποκοιήματα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να φωτιστούν λιγάκι απλετότερα. Έχουμε μια μακροπρόθεσμη δημοσιονομική προοπτική, αλλά έχουμε τώρα και τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματαγορές και στην πραγματική αγορά η πολιτική παροχής ρευστότητας δεν λειτουργεί, υπάρχουν κρατικές επενδύσεις για την αναζωγόνηση της οικονομίας και τίθεται το ερώτημα σε τι μπορεί να συμβάλλει η περιφερειακή πολιτική. με μια ταχύτερη παραδείγματος χάρη εφαρμογή μέτρων, με το να προταχθούν μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις οικονομικές δυνατότητες της περιοχές. Οπότε μετατοπίζεται η εστίαση της ε, περιφερειακής πολιτικής από μια βοήθεια από των ασθενεστέρων σε μια τόνωση της πολιτικής ε, ανάπτυξης, μάλλον δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε μια σταθεροποίηση της οικονομίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει <clears throat> να σκεφτούμε το αν θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες, πώς θα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τα συμπληρωματικά μέτρα και το κατά πόσο είναι απαραίτητη πλέον η, χρηματο... συγχρηματοδότηση. Εάν δεν χρειαζόμαστε καμία αλλαγή τα επόμενα 20 χρόνια στους κανόνες, τότε η συγχρηματοδότηση εξασφαλίζει ότι υπάρχει και η συνεισφορά των περιφερειών και των κρατών και δεν γίνονται επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν νόημα. Δεν, μπορούμε να, δεν γίνονται έτσι λοιπόν λαθασμένες επενδύσεις. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε είναι αν τώρα έχουμε προβλήματα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο για να εξασφαλίσουμε τη συγχρηματοδότηση, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δοθούν κάποια, κάποιες διευκολύνσεις πιστώσεων προς τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες, αλλά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, για ένα χρόνο ή κάτι τέτοιο, για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Όχι λοιπόν να άρουμε την υποχρέωση Τη ε, της Αλλά αν θέλουμε να βοηθήσουμε, να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να δράσουμε τώρα και αυτό σημαίνει να υπάρχει κάποια διευκόλυνση για τα κρατη Λοιπόν, έχετε κάποια τέτοια ιδέα στο μυαλό της να δώσετε τέτοιες σύντομες διευκολύνσεις, εξαμηνίες, έξι μηνών ενό χρόνου, ώστε τα χρήματα να μπορέσουν να αρεύσουν και να εκταμιευτούν με μεγάλη ταχύτητα, χωρί αυτό να σημαίνει μια αλλαγή κανόνα που μπορεί να χρονοτριβήσει. Ευχαριστώ πολύ, ο Γενικό ε, Διευθυντή. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Υπάρχουν ε, δύο ε, ειδών διευκολύνσεις. Της πρώτης μορφής ε, είναι οι προκαταβολές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν λειτουργικά ταμεία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Τα περισσότερα κράτη-μέλη άλλωστε χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά το 2009 για αυτό το σκοπό ε, βάσει της ε, έρευνας που κάναμε. Η άλλη περίπτωση είναι ε, η περίπτωση του IB. Δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη μέσω του IB να διευκολυνθούν και κατά την άποψή μας πρόκειται για κάτι ελκυστικό γιατί δίνει μια πιστοτική διευκόλυνση ε, με ε, την ασφάλεια των διευθυντικών ε, πόρων και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου καλά. Και νομίζω ότι αν συνδυάσουμε τις προκαταβολές και την πιστοτική διευκόλυνση, ε, τότε τα πράγματα είναι αρκετά ικανοποιητικά, γιατί δεν είχαμε καμία αντίδραση ε, όσον αφορά τα θέματα αυτά. Εγώ ε, ο ίδιος απέστειλα μόνο μια-δυο επιστολές σχετικά με κάποιες αμφιβολίες που είχαμε όσον αφορά την χρήση των προκαταβολών ε, και μελετούμε το ζήτημα αυτό, αλλά ε, το συνόλο δεν μπορώ να πω ότι υπήρξαν προβληματισμοί και επί της ουσίας δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να φανταστεί τα ιδιωτικά ταμεία χωρίς ε, συγχρηματοδότηση. Οπωσδήποτε πρόκειται για μία αρχή η οποία θα διατηρηθεί πέρα από οποιαδήποτε κυκλικά προγράμματα μπορεί να υπάρξουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ντελή και θα είναι ε, και θα έχουμε ακόμα μια ομιλήτρια και θα κλείσει ο κατάλογος των αφορετών. Κυρία Ντελή, καλημέρα κύριε Γενική Διευθυντά, καλώς ήρθατε. θα ακολουθήσω λίγο τη σκέψη του κυρίου Όλμπραϊτ. Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στη Γαλλία, αλλά να σας πω ότι η Γαλλία χρησιμοποίησε τα χρήματα για, την, ε, ε, για στεγαστικά προγράμματα. Πρώτον, γιατί δεν ζητήθηκε οποιαδήποτε τροποποίηση των λειτουργικών προγραμμάτων. Δεύτερον, γιατί κινητοποιήθηκαν οι ε, οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με τα προγράμματα στέγασης. Και τρίτον, γιατί υπήρξαν και εθνικά προγράμματα, όπως ας πούμε δάνεια για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Γιατί, γιατί δεν λαμβάνονται λοιπόν άμεσα μέτρα. Ας πούμε ένα άμεσο μέτρο θα ήταν να ξανανοίξουν άμεσα τα λειτουργικά προγράμματα και ε, να χρησιμοποιηθούν άμεσα οι πόροι μέχρι το 2013 έτσι ώστε να ε, ωφεληθούν όλοι από τα κονδύλια αυτά. Γιατί σήμερα δεν δίνεται μια απλή τεχνική συμβουλή έτσι ώστε και άλλα κράτη-μέλη να υποφεληθούν και να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστούμε. Κυρία Ιάννη, παρακαλώ. Όσον αφορά αυτό που είπατε, ναι, προφανώς. Μάλλον να το θέσω αλλιώς, λέει ο κύριος Άνε. Είναι γεγονός ότι το 2009 είμαστε λίγο διστακτικοί να καλέσουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να ανοίξουν τα προγράμματά τους διότι υπάρχει μία τάση στα ε, κράτη-μέλη όταν ανοίγουμε ένα πρόγραμμα και όταν το τροποποιούμε βλέπουμε ότι τα κράτη και οι περιφέρειες περιμένουν λίγο ε, να προσαρμοστούν στην αλλαγή και μετά να δουλέψουν πάνω στην αλλαγή πέρα από κάποιες επίγουσες περιπτώσεις θεωρήσαμε ότι το 2009 ήταν σημαντικό τα προγράμματα τα οποία είχαν εγκριθεί να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν και νομίζω ότι αυτό συνέβη στις περισσότερες χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Γαλλίας. Είχαμε καλό ποσοστό υλοποίησης. Τώρα, όπως είναι φυσικό, φτάνουμε στο μέσον ε, του χρόνου για τα ε, διαφορετικά ταμεία και επομένως ζητούμε ε, όλο και περισσότερο από τις περιφέρειες να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους. Συζητούμε λοιπόν με τις περιφέρειες και βεβαίως τους δίνουμε την δυνατότητα αυτή. Και κυρίως εάν υπάρχουν και άλλες επενδύσεις ε, στις οποίες ε, οι περιφέρειες ας πούμε είχαν βασιστεί και οι οποίες τελικά ε, δεν υλοποιούνται ας πούμε κάποιες αργοπορίες όσον αφορά επενδυτικά προγράμματα επιχειρήσεων. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες, κυρίως μεταξύ των παλαιών χωρών, που έχουν ήδη εθνικά προγράμματα που λειτουργούν καλά και καμιά φορά μπορεί να πούνε δεν χρειαζόμαστε τώρα για τα θέματα αυτά επί των οποίων εμείς ήδη εργαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε ε, και κοινοτικά κονδύλια. Ναι, βεβαίως, βεβαίως εμείς ε, συμβουλεύουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες όσον αφορά το τι γίνεται με τα προγράμματα. Αυτό που δεν κάνουμε, γιατί νομίζω ότι και εδώ είναι θέμα εταιρική σχέσης, αυτό που δεν κάνουμε λοιπόν είναι ε, δεν δίνουμε ε, οδηγίες, δεν επιβάλλουμε, δεν λέμε θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Οι δυνατότητες υπάρχουν, είναι ελκυστικές κατά την άποψή μου, πολλό δε μάλλον ε, όταν τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζει προβλήματα, ενδεχομένως λόγω της κρίσης, ε, αντιμετωπίζει προβλήματα στην υλοποίηση του συνόλου του αρχικού προγραμματισμού. Ε, ε, μου θέσατε και άλλο ερώτημα. Όχι, όχι, πολύ ωραία. Very much indeed, and I'd like to give the Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπριάν Ποκονέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ. Στην Επιτροπή μας, δύο μοναχα στοιχεία σε σχέση με την δράση των κρατών μελών στο Ευρώπη στα ευρωπαϊκά αυτά θέματα. Εμείς μπορούμε να αμοιβεοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό. Ότι μια περιοχή η οποία δεν καταναλώνει καλά τα ποσά της μπορούμε να τα μεταφέρουμε τα ποσά αυτά προς μια περιοχή η οποία καταναλώνει καλά τα ποσά αυτά. Αυτό θα βελτίωνε την, την εκταμίευση των ε, ποσών αυτών και θα και θα αξιοποιούσε ιδιαίτερα τη δράση αυτών οι οποίοι με τρόπο δυναμικό και θετικό κάνουν αυτές τις ενέργειες. Δεν ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Και τώρα κάτι πιο συγκεκριμένο. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί για μία πρωτοβουλία που λεγόταν ο έρασμος των τοπικά εκλεγμένων. Επιτρέπουν αυτή η πρωτοβουλία στους εκλεγμένους, στους τοπικούς, να γνωρίσουν άλλους τόπους και άλλες χώρες εκτός από τη δική τους. Είχε προετοιμαστεί μια γραμμή προϋπολογισμού για το 2009 για να προετοιμαστεί αυτή η διαδικασία. Πόσο, σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε λειτουργία αυτή η πρωτοβουλία. Εμείς στη Γαλλία είχαμε πάρει αιτήσει των τοπικό εκλεγμένο για αυτή την πρωτοβουλία. Τι να τους απαντήσω όταν με ρωτάνε. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Αν έρχεται το λόγο. Δύσκολο το ερώτημά σας. Για το πρώτο σας ερώτημα, εγώ πρέπει να πω, δεν έχω καταφέρει να σας εξηγήσω τα τεκτενόμενα με την κατάσταση νησιν 2. Στο τέλος του 2009, εμείς είχαμε σχετικά λίγα προβλήματα στο νησιν 2. και κυρίως επικεντρωμένα στην, σε μία χώρα μοναχα. Όχι, σε δύο χώρες, συγγνώμη. Σας είπα τα μισά μοναχα. Στην Ισπανία και την Ιταλία, όπου αναγκαστήκαμε να μπούμε τώρα σε μια διαδικασία, όπως ξέρετε, αλλά για το έτος 2007 υπάρχει μια πρόταση <clears throat> από την Κομισιόν, μια πρόταση επιτραπέζια πλέον, και η οποία προτείνει να βάλουμε το 2007 και το 2008 μαζί, κάτι το οποίο σημαίνει Νομίζω ότι υπάρχουν τα προβλήματα αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να εθνικοποιήσουμε την διαδικασία αυτή. Να θέσουμε το ερώτημα του αν θα πρέπει να προωθήσουμε τον κανόνα αυτό και να φτάσουμε στο νησιν 3 και όχι μόνο στο νησιν 2. Και να δούμε αν πρέπει να έχουμε ένα νησιν τρία και όχι νησιν δύο μονάχα για να εξασφαλίσουμε ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν αργά να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ή θέλουμε να διατηρήσουμε εδώ την ε, απειλή αυτή του να χαθούν τα λεφτά που κατά κάποιο τρόπο προωθεί τις προσπάθειες σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό είναι μια πραγματική πολιτική επιλογή γιατί πρέπει να είμαστε σαφείς. Το νησιν 2 δεν έχει καμία επιστημονική βάση για να φτάσουμε να λέμε ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. και ούτως ή άλλως το είναι πολύ πιο δύσκολο για τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας όταν υπάρχουν πολλές χώρες διαμεθοριακές με διαφορετικές κουλτούρες από ό,τι στην περίπτωση του προγράμματος mainstream. Και εκεί υπάρχουν πάλι κάποιες δυσκολίες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν για το μέλλον και η πρότασή σας είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Για τον έρασμο των τοπικά εκλεγμένων. Δεν ξέρω αν ο Χουάν μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ξέρω ότι έχουμε κάνει κάποιες μελέτες για τα θέματα αυτά. Εγώ ήμουν πολύ υπέρ αυτό των μέτρων στην αρχή, αλλά κατανόησα ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα που προέρχονται από την δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα, αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμαστε και για να σας δώσω πιο ενδελεχείς πληροφορίες θα πληροφορηθώ και θα σας δώσω και μια έγγραφη απάντηση. Αλλά όλα τα προπαρασκευαστικά σχέδια και, και τα πιλωτικά σχέδια ήταν από τα πιο δύσκολα που χρειάζεται να κάνουμε σε τεχνικό επίπεδο. Γιατί σε επίπεδο διοικητικό, δεν έχουμε τις απαραίτητες δομές, όπως για τον έρασμο των φοιτητών, όταν είναι μια υπόθεση μεταξύ πανεπιστημίων, που μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση. Η ιδέα παραμένει όμως μια έγκυρη ιδέα και πρέπει να τη δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γενικέ Διευθυντά για τα στοιχεία, τους αριθμούς και τα, τη ζήτηση που είχαμε και πραγματικά περιμένουμε με ανυπομονησία την προσεχή μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ επίσης πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά που είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, ε, Ολενίτσακ είναι εδώ, θα του δώσω το λόγο. Θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση που έχει προετοιμάσει ο κύριος Ολενίτσακ σχετικά με την στρατηγική για τη Βαλτική και το ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχή. Δεν θα πάρουμε καμία απόφαση σήμερα. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Ολενίτσακ, έχετε το λόγο. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić dokument roboczy w sprawie strategii Unii Europejskiej dla ναι, θα αναφερθώ στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής, καθώς και για το ρόλο που θα παίξουν μακροπεριφέρειες στη μελλοντική πολιτική συνοχή. Η στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα είναι η πρώτη μέχρι στιγμή περιεκτική κοινή στρατηγική για τις μακροπεριφέρειες. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο η στρατηγική της Βαλτική θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια στρατηγική πιλωτικού χαρακτήρα και τα συμπεράσματα τα οποία θα εξαχθούν από την εφαρμογή της θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη περαιτέρω στρατηγικών για τις ευρωπαϊκές μακροπεριφέρειες. Αυτή η στρατηγική υιοθετήθηκε ακολουθώντας πλατιές διαβουλεύσεις όχι μόνο με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά επίσης και με πανεπιστήμια, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος. Το γεγονό ότι πάρα πολλές ομάδες συμμετείχαν στο σχέδιο προγράμματος. Η στρατηγική βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες όσον αφορά την πιο αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων, δηλαδή προστασία του περιβάλλοντος, ούτω ώστε να βελτιθεί η προσβασιμότητα των ε, περιοχών και να αυξηθεί η ασφάλεια. Πέρα από αυτούς του τέσσερι τομέί, του μελλοντικά, θα πρέπει να εξετάσουμε ένα άλλο τομέα που αφορά τα, την κοινωνική και ακαδημαϊκή πτυχή σε σχέση με τι καινοτομίε. Η στρατηγική και τι μακροπεριφέρειες θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να επηρεάσει την ε, μεγαλύτερη ε, ολοκλήρωση πολιτών και κοινωνία σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Τα σημεία κίνησης για τη στρατηγική στις, ε, βασίζονται στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες για τις ε, περιφέρειες τόσο όσον αφορά τις ε, διμερείς συνεργασίες μεταξύ των χωρών και τη συνεργασία μεταξύ χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Βαλτική. Καταρχήν θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια στρατηγική για την Βαλτική και να ορίσουμε κάποιους στόχους που θα πρέπει να εκπληρωθούν από κοινού και στη συνέχεια θα πρέπει να εγκριθούν κάποια προγράμματα ούτω ώστε ε, να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι. Μία άλλη βασική αρχή για τη χάραξη στρατηγική είναι μια συντονισμένη στρατηγική για ε, συντονισμένε δράσει που να περιλαμβάνουν όλου του στόχου. Σήμερα οι στόχοι για την Βαλτική για τη στρατηγική τη Βαλτική, εφαρμόζονται κυρίω χρησιμοποιώντα τα ταμεία πολιτική συνοχή. Αλλά μελλοντικά και, άλλες, και άλλοι τομεί θα πρέπει να επικεντρωθούν στη στρατηγική για αυτή την περιοχή και θα πρέπει να περιλαμβάνουν κυρίως την κοινή γεωργική πολιτική, την πολιτική αλίας, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη. Η στρατηγική προβλέπει μια στενότερη συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οποίων οι επικράτειες εμπίπτουν στη λειτουργική, στο λειτουργικό τομέα των μακροπεριφερειών, είτε επειδή έχουν μια επίδραση στις μακροπεριφέρειες. Στα δική εμπίπτωση αρμοδιότητων χωρών μελών, οι δραστηριότητε συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονό ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επαρκεί ε, πόρου, ούτε χρηματοοικονομικού, ούτε ανθρώπινου πόρου, ούτε ώστε να μπορέσει αποτελεσματικά να αποπτεύσει την εφαρμογή αυτή τη στρατηγική. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η, η έκθεση εφαρμογή τη στρατηγική που θα παρουσιαστεί το 2011 να παρουσιάζει επακριβώ τα συμπεράσματα και να παρέχει τη βάση το για βελτίωση. Κατά τη διάρκεια της ε, Πολωνικής Προεδρίας εκεί θα πρέπει να βελτιωθεί για το μέλλον. Ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Καταρχήν θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα κοινωνικά συστήματα και τι ε, οικονομίες ούτως ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει από πιο προηγμένες χώρες, όπως είναι οι, χώρες της, οι χώρες. Αυτά τα παραδείγματα θα μπορούσαν να εξοπιθούν από άλλες χώρες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες και που δαπανούν <coughs> λιγότερα κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις προκλήσεις κλειδί για το μέλλον. Επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα στην περιοχή. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι ο πληθυσμός γυράσκει σε αυτές τις μακροπεριφέρειες. Η ανάπτυξη θα πρέπει να παραμείνει η μεγαλύτερη μίσον προτεραιότητα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική βεβαίω και ένα ιδιαίτερο σημαντικό θέμα για το μέλλον είναι ο προπολογισμό χρηματοδότηση στρατηγική. Όπω είπα ήδη, η στρατηγική για τη Βαλτική αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια εφαρμογή ενό υφιστάμενου προπολογισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή διακριτό προπολογισμό. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε κατά πόσο η στρατηγική για της μακροπεριφέρειας θα πρέπει να έχει ένα ξεχωριστό προπολογισμό που θα αφιερώνεται στον συντονισμό των δράσεων και επίσης ε, στην εφαρμογή των κοινών προγραμμάτων. Αυτό το ερώτημα δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, παραμένει ανοιχτό. Μια σημαντική πρόκληση που συνδέεται με την εφαρμογή της στρατηγικής και η οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς είναι τα θέματα μεταφοράς. Πλωτές μεταφορές, αλλά και σιδηροδρομικές μεταφορές, οδικές μεταφορές στην περιοχή της Βαλτικής. Επίσης έχουμε θέματα που συνδέονται με την ενέργεια και θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονό ότι ο βόρειος αγωγός ε, δεν βρίσκεται σε υποθετική φάση αλλά είναι υφίστατος οντότητα και δεν θα πρέπει να θέτουμε το ερώτημα κατά πόσο θα κατασκευαστεί. Είναι σίγουρο ότι θα κατασκευαστεί. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τις συνέπειες που θα έχει για την οικονομία αλλά και την ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις όσον αφορά τις μεταφορές και την προσβασιμότητα των λιμένων ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα με ενεργειακούς όρους και όρους οικονομίας είναι η της Βαλτικής είναι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών στη Βαλτική. Ε, η χρήση ολόκληρης της περιοχής, για παράδειγμα, για την ε, παραγωγή βιομάζας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, για ενεργειακούς σκοπούς. Ένα άλλο θέμα ζωτικής σημασίας είναι η εμβέλεια της μακροπεριφέρειας. Οι μακροφέρειες θα πρέπει να καλύπτουν μόνο αυτούς τους τομείς που έχουν οριστεί επακριβώς ή θα πρέπει να ερμηνεύονται οι μακροπεριφέρειες με έναν πλατύτερο τρόπο. Γιατί οι στόχοι που θέλουμε να εφαρμόσουμε εντός της περιοχής αυτές, αυτής, έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από τα σύνορα της ε, λόγω μακροπεριφέρειας, για παράδειγμα, όσον αφορά τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και σε ορισμένε περιπτώσεις καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας των χωρών μελών. Και όταν μιλούμε για τη Βαλτική θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με τα ποτάμια ε, ε, που είναι σε χώρες εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκβάλλουν στη Βαλτική. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τις συνέπειε και τα συμπεράσματα της εφαρμογής στρατηγικής για την Βαλτική θάλασσα και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτή την εμπειρία. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα όσον αφορά την ε, στρατηγική για την για αυτή τη μακροπεριφέρεια. Θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται με τις άλλες ε, μακροπεριφέρειες, ούτως ώστε να χαράξουμε μια νέα πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, ο οποίος προετοίμασε αυτό το έγγραφο εργασίας και μας έκανε και μια προφορική παρουσίαση η οποία συμπλήρωσε το εγγραφό του. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα καλό θεμέλιο για την περαιτέρω επεξεργασία από την Επιτροπή μας και για να μπορέσουμε να θέσουμε τα ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την στρατηγική της Βαλτικής. Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι η Βαλτική βρισκόταν πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα στο παρελθόν <clears throat> και είχε επηρεαστεί από την διέρεση της Ευρώπης σε ανατολική και δημοκρατική και ότι πριν από 20 χρόνια ακόμα βρισκόταν σε ένα δικτατορικό καθεστώς. Αυτά είναι τα στοιχεία του παρελθόντος, το οποίο είναι σχεδόν νοπό ακόμα αυτό το οποίο είναι σημαντικό όμως είναι ότι η Βαλτική έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς, την, ε, τα βόρεια και τα ανατολικά και τώρα η Βαλτική είναι μια εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συνδέει τους λαούς και τα κράτη της περιοχής και φυσικά αποτελεί μια πρόκληση για μας υπό την έποψη της περιφερικής πολιτικής πώς θα αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά προβλήματα, τα προβλήματα του περιβάλλοντος, τις ε, συγκοινωνιακές συνθέσεις, τα κοινωνικά θέματα, πώς θα επιλύσουμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα και ήδη μας έχει κάνει μια εισαγωγή στην προβληματική αυτή ο εισηγητής. <clears throat> Υπάρχουν ε, και υψηλού, υψηλές προσδοκίες από όλους τους εμπλεκόμενους, τους κατοίκους της περιοχής γύρω από την Βαλτική θάλασσα και των κρατών μελών. Αυτά είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζει όχι μονάχα η Κομισιόν, αλλά και το Κοινοβούλιο και υπάρχουν και κοινά προγράμματα και σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί από τους εταίρους οι οποίοι εμπλέκονται στην Βαλτική, ώστε να υπάρξει μια κοινή ε, περιφερειακή προβληματική σε σχέση με την Βαλτική. Ο κύριος Ολενίτσακακ το τόνισε και αυτό προηγουμένως. Εμείς με την στατική της Βαλτικής για πρώτη φορά ξεκινούμε μια αντιμετώπιση σε επίπεδο μακροπεριφέρειας και γνωρίζουμε ότι επίκειται μια τέτοια αντιμετώπιση και για την περιοχή του Δούναβη. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον της πολιτικής συνοχής γιατί συνδυάζονται με μια τέτοια πολιτική όλα τα ζητήματα των μακροπεριφερειών. Επομένω, δεν πρέπει να δούμε την πολιτική τη Βαλτική μονάχα μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική λόγω των προβλημάτων τα οποία συνάπτονται με την περιοχή τη Βαλτική και επίση θα πρέπει να υπάρξει και η απαραίτητη πολιτική από τα κράτη-μέλη <clears throat> να συμμετέχουν σε αυτέ τι ε, διαδικασίε. Η γερμανική Bundestag πριν από τις εκλογές είχε πάρει μια απόφαση ότι και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα πρέπει και αυτή να συμμετάσχει στα τεκτενόμενα στον χώρο της Βαλτικής. Ο κύριος Όλινετσάκ έθεσε ορισμένα ερωτήματα στα οποία θέλω να αναφερθώ και εγώ. Το θέμα της συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να το λησμονήσουμε. Η στρατηγική μας θα έχει νόημα μονάχα εάν μπορέσει να συμπεριλάβει και τη Ρωσία. Γνωρίζουμε ότι πολλά, πολλά, πολλά, από τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ε, ε, Βαλτική δεν είναι τοπικά προβλήματα, είναι προβλήματα τα οποία προέρχονται και από βαθύτερα στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συζήτηση και με την Ρωσία, να έχουμε μια αντιπροσωπεία της Δούμα, της Ρωσικής Δούμα και να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό μέσα στη μεικτή την... Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασία με τη Ρωσία και να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα την προβληματική που έχει να κάνει με το ρόλο τη Ρωσία στη Βαλτική. Επίση, τα χρηματοοικονομικά θέματα τα ανέφερε ο εισηγητή σα. Έχουν θεσπιστεί τα λειτουργικά προβλήματα για αυτή τη χρονική περίοδο και όταν δούμε τα προγράμματα αυτά τα οποία έχουν ε, ήδη <clears throat> διατυπωθεί και ζητηθούν πρόσθετα κονδύλια ή όταν έχουμε να εκπονήσουμε νέα σχέδια εξ αρχής, τότε θα πρέπει όλη αυτή η στοχοθεσία που αναφέρθηκε από τον εισηγητή να είναι το κεντρικό σημείο, να είναι το κέντρο βάρους. Επίσης χαίρομαι για το γεγονός ότι ο εισηγητής τόνισε ότι αν επιτυχείς η στρατηγική της ε, Βαλτικής δεν θα είναι μονάχα ένα θετικό στοιχείο σε επίπεδο ενιολογικό, αλλά θα πρέπει να έχει και μια υλική πλευρά η οποία να είναι επιτυχής. Και αναφέρθηκε και το θέμα του Nord Stream, του αγωγού που θα περάσει στη Βαλτική. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι σε πολλές συζητήσεις οι οποίες αφορούν τη στρατηγική της Βαλτικής έρχεται σαν αντανακλαστικό και η συζήτηση για το North Stream. Εγώ νομίζω ότι είναι βέβαια ευρύτερη η στρατηγική της Βαλτικής από μόνο η συζήτηση η οποία έχει πάρει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το North Stream και επομένως το σχέδιο αυτό προφανώς θα πρέπει να παίξει ένα θετικό ρόλο για την περιοχή αυτή, να μην αντιμετωπιστεί μονάχα σαν μια διμερής υπόθεση, αλλά κάτι που ενδιαφέρει το σύνολο χώρο της Βαλτικής και επίσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να το συζητήσουμε. <clears throat> και κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό, το τελευταίο ερώτημα το οποίο έθεσε ο εισηγητής, αν οι μακροπεριφέρειες είναι πραγματικά λειτουργικές μονάδες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να λύσουν τα προβλήματά μας και αν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επωφελώς τις προκλήσεις της πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι αυτό είναι πράγματι ένα εύστοχο ερώτημα το οποίο θέτει ο εισηγητής και ε, γύρω από αυτό το θέμα θα πρέπει να περιστραφεί η περαιτέρω προβληματική μας για τη στρατηγική της συνοχής και χαίρομαι για την ευκαιρία που θα έχει ο εισηγητής με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές να επεξεργαστεί περαιτέρω το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσέλερ για την πλήρη σας παρέμβαση και δήλωση. Ο Γιάνν Όλμπρεχτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα είμαι πολύ πιο σκεπτικιστής σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Γιατί κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το θέμα του Δουνάβεως υπήρξαν ορισμένα θέματα πολύ σημαντικά τα οποία συζητήθηκαν. Και θα ήθελα να τα πω αυτά και στον κύριο Λενίτσεκ γιατί με τρόπο πάρα πολύ σαφή απαντά στις ερωτήσεις ε, οι οποίες τίθενται. τίθενται. Βεβαίως, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι θα πρέπει να προωθηθούν ευρείας κλίμακος λύσεις. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως ε, και στην περιφέρεια της Βαλτικής και του Δούναβη και στην Μεσόγειο ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ευρωπαϊκή στρατηγική, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χώρες ε, οι οποίες έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τις περιφέρειές τους το ίδιο ισχύει και για τη Βαλτική, το ίδιο ισχύει και ε, για τον ε, Δούναβη. Και στα πλαίσια ε, της διαδικασίας 2020 οι χώρες της Βαλτικής βεβαίως αποτελούν προτεραιότητα. Τώρα το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να ε, προχωρήσουμε ε, σε προγράμματα σωστά, γιατί διαφορετικά ε, θα πρόκειται για μια απλή περιγραφή πολυμερών σχέσεων. Το ίδιο ισχύει και για τη στρατηγική για την περιφέρεια του Δουνάβεως. Καλό είναι να λέμε ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κρατών μερών, αλλά, ε, μελών, αλλά βεβαίως ε, δεν μπορεί να είναι και περιορισμένος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βελτιωθούν ακόμα και οι πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης η στρατηγική υλοποίηση θα πρέπει να φέρει το στίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και εάν πρέπει να προχωρήσουμε σε λειτουργικές και μακροπεριφέρειες θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε την φιλοσοφία των πληρωμών. Ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στις μακροπεριφέρειες αλλά εάν δεν το κάνουν τότε δεν θα λειτουργήσει καλά το, το σύστημα νομίζω ότι δεν μπορεί μονάχα από τα εθνικά πακέτα να προχωράει να ε, εκπορεύεται η χρηματοδότηση. Ζητήσαμε Ρωτήσαμε μάλλον την ε, μέλουσα επίτροπο εάν συμφωνούσε με μία πρόσθετη γραμμή του προπολογισμού και απάντησε αρνητικά ότι δεν ε, θέλει αυτήν την ε, επιπρόσθετη γραμμή του προπολογισμού και επομένως θα πρέπει να αποφασίσουμε είτε θα αλλάξουμε την προσέγγιση από τα εθνικά πακέτα προς τις μακροπεριφέρειες ή θα πρέπει να βρούμε επιπλέον κονδύλια ή θα πούμε ότι η περιφέρεια της Βαλτικής ε, θα πρέπει να μπει στον στόχο 3 και θα πρέπει να αλλάξουν βεβαίως ε, και τα ποσοστά γιατί διαφορετικά δεν έχει έννοια. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι ο κύριος Ολενίτσακ ε, ανεφέρθη σε πολύ ευαίσθητα θέματα γιατί δεν είναι μονάχα θέμα στρατηγικής συνοχής αλλά οτιδήποτε αυτή συνεπάγεται. Και βεβαίως ε, ε, εφαρμο... άπτεται πολλών πολιτικών. Γι' αυτό νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να τροποποιήσουμε την πολιτική συνοχής με την πολιτική στη Βαλτική. Γιατί αλλιώ οι ιδέε όπω αυτή, οι στρατηγικέ όπω αυτή θα παραμείνουν σε ένα συμβολικό επίπεδο. Απλώ θα σημαίνει ότι μερικά κράτη-μέλη θα κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και θα συζητούν, αλλά αυτό δεν θα μπορέσει να αποτελέσει μια πραγματική στρατηγική, αν μείνει μονάχα σε ένα συμβολικό επίπεδο. Όταν συζητήθηκε η πολιτική για το Δούναβι, Υπήρξαν πολλοί βουλευτέ οι οποίοι είπαν ότι θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν ειδικά κονδύλια για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολιτική. Είναι ειδικέ πολιτικέ οι οποίε πραγματικά έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν την εδαφική συνοχή. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνήσουμε. Από την άποψη αυτή, τα πιλωτικά σχέδια θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια διαφορετική μεθοδολογία. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, <clears throat> όταν δεν υπάρχει μια συνοχή πολιτικών, όσο και αν σκεφτόμαστε για τις μακροπεριφέρειες, όλα αυτά παραμένουν στον αέρα. <clears throat> Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι να υπάρξει μια πραγματική χρηματοδότηση των σχεδίων που υποστηρίζουν τι μακροπεριφέρειες. Και μέσα στα πλαίσια τη στρατηγική Λισαβόνα θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για όλε αυτέ τι χώρε και τι περιφέρειες. Και είναι γεγονό ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει ευκαιρίε σε σχέση με τη στρατηγική τη Βαλτική. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μιλάει για την περιοχή της Βαλτικής. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος. Κυρία Μάνερ, σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής <clears throat> έχει κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Νομίζω ότι περιλαμβάνει η παρέμβασή του φιλόδοξους στόχους με τους οποίους συμφωνώ και θέλω να ευχαριστώ και τη Γραμματεία για τη συνεργασία τους. <clears throat> Όσο εξετάζουμε αυτό το έγγραφο για τη στρατηγική της Βαλτικής και τις αρχές που πρέπει να τη διέπουν, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή η στρατηγική να μην καλύπτει μονάχα τη Βαλτική, αλλά και την σύνολη περιοχή γύρω από τη Βαλτική. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση όχι μόνο στις παράκτιες περιοχές και τις πόλεις που είναι κοντά σε θάλ, στη Βαλτική, αλλά την εσωχώρα, την ενδοχώρα μάλλον της Βαλτικής που είναι πολύ σημαντική, ιδίω όταν μιλάμε για εσωτερικούς υδάτινους δρόμους και τις δυνατότητες που παρέχουν αυτές οι εσωτερικές υδάτινες οδοί σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο 4 στο έγγραφο του εισηγητή, όπου αναφέρονται οι μελλοντικέ προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο πρώτο αυτό τμήμα <clears throat> υπάρχει μια σαφής διάκριση η οποία γίνεται μεταξύ των παλιών και των καινούριων κρατών μελών. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα πρέπει επιτέλους να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από μια τέτοια τυπολογία. Θα ήθελα τα κρατημέλη να μην κατηγοριοποιούνται με ένα τέτοιο τρόπο. Πιστεύω ότι θα ήταν πιο πρόσφορο να μιλάμε για το δυναμικό της κάθε περιφέρειας και πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο, ιδίως σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την τεχνογνωσία. Και θα εφιστούσα ιδιαίτερα την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο στόχος αυτός <clears throat> δεν εξαρτάται μονάχα από το ΑΕΠ όταν μιλάμε για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία. Θα πρέπει να ληφθούν εδώ οι διαφορές, οι διαφορές επίπεδου ανάπτυξης και επίσης οι διαφορές οι οποίες ενυπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος και όχι μονάχα οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά στις μελλοντικέ λοιπόν προκλήσεις, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις καθαρές τεχνολογίες, <clears throat> στους τρόπους με τους οποίους τα κράτη-μέλη μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη καθαρών λύσεων για το περιβάλλον, αλλά αυτό είναι και σημαντικό για την ανάπτυξη της οικονομίας. Σε επίπεδο στρατηγικής λοιπόν, <clears throat> η ανταγωνιστικότητα της περιοχής θα πρέπει να είναι μία από τις κύριες μέρημνές μας. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε τις προκλήσεις οι οποίες αφορούν την δημογραφική γύρανση και επίσης να δώσουμε την απαραίτητη έμφαση στα θέματα μεταφορών, ιδίως οι μεταφορές με εσωτερικούς υδάτινους δρόμους. Επίσης, σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας, αντιμετωπίζεται πολύ σωστά από τον εισηγητή. Θα ήταν χρήσιμο όμως να έχουμε μια πιο εκτενή αναφορά για τα ενεργειακά ζητήματα. Εάν θέλουμε εμείς να λάβουμε υπόψη μας και να εκμεταλλευτούμε τις ανανεώσιμες ενέργειες, υπάρχει μια πλειάδα δυνατοτήτων για έρευνα και ανάπτυξη στην περιοχή της Βαλτικής. Και αναφέρεται στο έγγραφο του εισηγητή η αιωλική ενέργεια <clears throat> και χαίρομαι που ο εισηγητής αναφέρεται επίσης και στην εκμετάλλευση της βιομάζας γιατί έχουμε πολλά πολλά πολλά δάση στην περιοχή αυτή κάτι το οποίο μπορεί να είναι μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για τον ενεργειακό τομέα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης το θέμα του ρόλου των τρίτων χωρών. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω το έχετε αντιμετωπίσει κύριε Σιγητά πολύ ωραία στο εγγραφό σας, ιδίως όταν αναφέρεστε στα ωφέλη τα οποία μπορούμε να προσποριστούμε μέσω της καλύτερης προσβασιμότητος και της ανάπτυξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές και της καλύτερης συνεργασίας με όμορες χώρες. Για τη χρηματοδότηση. Επειδή είναι παρόν και εκπρόσωπος της Κομισιόν, θα ήθελα να ρωτήσω <clears throat> ποιος είναι ο στόχος της Κομισιόν πώς θέλει να αντιμετωπίσει αυτά τα 20 εκατομμύρια, με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτήσουμε στο μέλλον και την, τις μακροπεριφέρειες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω πρώτον ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ε, συζητούμε, που ξεκινήσατε τη συζήτηση το θέμα αυτό και επίσης ε, χαίρομαι που οι υπεύθυνοι της Βαλτικής θάλασσας ε, ξεκίνησαν όλη αυτή τη διαδικασία για προγράμματα, για συνεργασία, δηλαδή μας δείχνουν το δρόμο για τον εξορθολογισμό των περιφερειακών πολιτικών στην Ευρώπη, πράγμα απολύτως απαραίτητο δεν μπορούμε να καταλάβουμε νομίζω αυτά τα αποθέματα ε, αποτελεσματικότητας τα οποία κρύβονται σε αυτές τις ε, προσεγγίσεις ε, συνεργασίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ και δύο μήνες ε, δεν μπορούμε να, δεν έχουμε καμία ναυτική ε, θαλάσσια διασύνδεση ανάμεσα στην Κορσική ε, και την Σαρδινία. Δηλαδή για να πάει ένα εμπόρευμα από την Κορσική στη Σαρδινία θα πρέπει να περάσει από την Κορσική στη Γαλλία, από τη Γαλλία οδικό στη Γένοβα και από τη Γένοβα ξανά με πλοίο στην Σαρδινία. Αυτό πραγματικά είναι απίστευτο, είναι παράλογο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να Πίσω με τις ε, περιφέρειες να σκεφτούν πραγματικά στα πλαίσια μακροπεριφέρειας για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Όμως θα ήθελα να πω ότι απογοητεύομαι από την ε, ε, Ισπανική Προεδρία η Σουηδική Προεδρία ήταν ε, πολύ δραστήρια σε σχέση με την Βαλτική. Ε, η, η Ουγγρική ε, είναι, φαίνεται, πολύ, θα είναι πολύ δραστήρια για τον Δούναβη, αλλά η Ισπανική δεν δείχνει καμία διάθεση να είναι δραστήρια όσον αφορά την Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε φαινό την εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα στη Βαλτική, να την ενδυναμώσουμε, να μας πει η Επιτροπή Επιτροπή τι ακριβώς προτίθεται να κάνει όσον αφορά ε, το δημοσιονομικό σχέδιο, όσον αφορά τον προπολογισμό έτσι ώστε να ε, παρακολουθούν περαιτέρω συνεργασίε και έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα τα προγράμματα. Τέλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει την ιδέα ε, ότι οι μακροπεριφερειακές συνεργασίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό άξονα, αποτελούν ένα αποθεματικό δυναμισμό που είναι σημαντικό για όλες τις περιφέρειες. Ένα λεπτό. Και όπως είπε και να μιλήσω και εγώ και ε, ε, όπως αναφέρθηκε και ο Φρανσουά ε, Αλφονσί, να μιλήσω και εγώ για την Μεσόγειο να πούμε ότι η περιφέρεια της ε, Μεσογείου ήταν μια διαδικασία top-down, τελείως διαφορετική, ενώ η, ε, η στρατηγική για τη Βαλτική και η στρατηγική για τον πύρο που ξεκινάει τώρα ήταν bottom-up ε, διαδικασία. Απολύτως μέσα στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής με στενή συνεργασία με, τη, με πολλές άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Επομένως ε, βασίζεται σε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και σίγουρα βασίζεται σε υφιστάμενες πολιτικές. Βεβαίω πρόκειται για πολιτική διεργασία, αλλά αυτή δεν, αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος. Για την Μεσογειακή Ένωση έχουμε διαφορετικές προσδοκίες αλλά βεβαίως αν θέλετε μπορούμε να δούμε εάν ε, θα έχουμε στο μέλλον και τη δυνατότητα να έχουμε, μια, ε, να έχουμε δημιουργία μακροπεριφέρειας και επομένως συγκεκριμένες μακροπολιτικές. Ε, so now the next speaker is Thomas Deutsch. Thomas Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να ε, συγχαρώ τον κύριο Ολένιτσακ για την εξαίρετη εργασία του. Κατά την άποψή μου, αυτό το έγγραφο εργασίας παρουσιάζει ένα εξαιρετικό στοιχείο. Δηλαδή, με εξαίρετο τρόπο ασχολείται με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ε, εν, ε, να εμβαθυνθούν. Ε, και συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και αυτά που είπε ο τελευταίος συνάδελφος που μίλησε. Λοιπόν, λέει ένα ρητό ότι σε κακές ερωτήσεις μονάχα κακές απαντήσεις μπορούν να δοθούν, αλλά εδώ γίνεται κι άλλο ένα λάθος. Εάν κάποιος κάνει ε, ένα σωστό ερώτημα και ο κύριος Ολένιτσακ έθεσε πολύ σωστά ερωτήματα. Ε, αυτά τα καλά ερωτήματα δεν απαντώνται σωστά. Εάν ε, λοιπόν δεν απαντήσουμε σωστά σε σωστές ερωτήσεις τότε κάνουμε ακριβώς το ίδιο λάθος όπως όταν απαντάμε άσχημα σε μια άσχημη ερώτηση. Ο κύριος Ολένιτσεκ μας έδωσε ένα εξαίρετο έγγραφο εργασίας και επομένως, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να ρωτάμε συνέχεια τα ίδια πράγματα, να θέτουμε διαρκώς τα ίδια ζητήματα, αλλά θα πρέπει πλέον να έρθει ο καιρός των απαντήσεων, να απαντήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, συγγνώμη, περιμένουμε απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και βεβαίω και από το Συμβούλιο, να μας πει τι συμβαίνει με το μέλλον της πολιτικής συνοχής και βεβαίως σε αυτά τα πλαίσια το ερώτημα του μέλλοντος των, ε, των μακροπεριοχών, των μακροπεριφερειών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην στήριξη και τη μη στήριξη. Ε, κοιτάξτε, εάν στηρίξουμε τις μακροπεριφέρειες ε, θα υπάρξουν και θα έχουν ένα σωστό μέλλον. Εάν δεν τις στηρίξουμε πάλι θα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά με ποιο τρόπο. Ε, δηλαδή, εάν δεν τη στηρίξουμε, θα τις αφήσουμε στο έλεος ε, των ε, συνθήκων και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη συμβολική σημασία η κίνηση που θα κάνουμε. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα σωστά ερωτήματα ε, και να δούμε τι ε, σωστές απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε στα ερωτήματα αυτά. Γιατί αν αφήσουμε τις περιφέρειες ε, στην τύχη τους, εντάξει, θα είναι περιφέρειες και όπως λέμε και στα Ουγγρικά, τι θα γίνει, ναι, θα βάλει η φοράδα Φερετζέ και τι σημαίνει, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, θα τις αφήσουμε στην τύχη τους. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα των ε, μακροπεριφερειών ε, με ε, τρόπο εμπνευσμένο κατά την άποψή, κατά την μου και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να πάρουμε πολύ σαφείς θέσεις. Εάν αποφασίσουμε ότι συμφωνούμε, ότι λέμε ναι, απαντάμε ναι στο ερώτημα ότι αν πρέπει να υπάρχουν μακροπεριφέρειες, τότε θα πρέπει να βάλουμε όλα τα δυνατά μας έτσι ώστε να τις χρηματοδοτήσουμε, να τις στηρίξουμε έτσι ώστε να έχουν δίπλα τους την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο ε, Συνοχής με βοήθεια είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα είτε από άλλους φορείς. Μα γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική γραμμή στον προϋπολογισμό που να αφορά ε, τις μακροπεριφέρειες. Αλλά είδαμε ότι οι Επίτροποι δεν συμφωνούν με αυτό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και άλλο ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο οργανισμός ο οποίος ε, θα ε, είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των μακροπεριφερειών. Έχουμε τη μακροπεριφέρεια της Βαλτικής, σχηματίζεται και η μακροπεριφέρεια του Δούναβη. Θα υπάρξουν και άλλες μακροπεριφέρειες Εάν όμως δεν υπάρξει συνολικός συντονισμός, τότε σίγουρα δεν πρόκειται να προχωρήσει καλά. Ε, θα πρέπει να υπάρξει εναρμονισμένη, συντονισμένη δράση. Τα πράγματα να γίνονται με τη σειρά τους και σωστά γιατί πολύ συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λειτουργούμε λίγο βάζοντας ε, το κάρο μπροστά από τα βόδια και επομένως το αποτέλεσμα είναι αντίθετο από αυτό που ε, το αρχικά. Τρίτο ζήτημα, η εφαρμογή πώς μπορούν να οριστούν αυτές οι μακροπεριφέρειες. Τώρα, στην ε, περίπτωση της Βαλτικής, ε, μιλάμε μόνο για τις παράκτιες περιοχές ή μήπως θα πρέπει να λάβουμε ε, και να συνυπολογίσουμε, να λάβουμε υπόψη μας και την ενδοχώρα. Να μιλήσουμε για, περισσότερο για λειτουργικές περιοχές. Υπάρχει κι άλλο ένα ερώτημα. Ποιο είναι το σύστημα αξιολόγησης των μακροπεριφερειών και αυτό τίθεται σαν ερώτημα στο έγγραφο εργασίας. δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ε, ένα νέο θεσμό στην περιφερειακή πολιτική για να δούμε, ε, να διαπιστώσουμε εκ των υστέρων ότι δεν μπορούμε να την ε, αξιολογήσουμε. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθεί και ένα σύστημα αξιολόγησης έτσι ώστε τα στοιχεία να είναι και συγκρίσιμα. Ακόμα και τα στοιχεία μεταξύ των μακροπεριφερειών να μπορεί να γίνει σύγκριση επί βασίμων στοιχείων ανάμεσα ας πούμε στη μακροπεριφέρεια της Βαλτικής και του Δούναβη. Αυτά. Voorzitter, dank u wel. Ook ik eh, dank voor, eh, voor de notitie. Ik Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν θα ήθελα να δυσχεράνω περαιτέρω την ε, κατάσταση. Απλώς ε, θα ήθελα να εμπλουτίσω λίγο τη συζήτηση. Εγώ έχω σπουδάσει βιοφυσική και μπορώ να σας πω ότι το, τα περιφερικά θέματα δεν πάβουν ποτέ. Ανεξάρτητα από επίκαιρα θέματα, θέματα συμμαχιών κλπ. Η συζήτηση για την περιφερειακή πολιτική δεν πάβει ποτέ. Και ε, το ζήτημα της μακροπεριφέρειας ανακύπτει και στο Συμβούλιο. Η σκέπ, οι οι προβληματισμοί συγγνώμη, σχετικά ε, δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 90. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν δύο παρατηρήσεις. Ναι, δεν θέλω να δυσχεράνω την κατάσταση, αλλά θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε μία έννοια, μία διευκρίνηση της έννοιας της περιφερειακής συνοχής. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερος σημαντικό όσον αφορά τη μακροπεριφέρεια γιατί τότε θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια διαφορετική αυτο ειναι ιδιαίτερο σημαντικο οσον αφορα τη μακροπεριφερεια γιατι γωνία για τι εξελίξει στην Ευρώπη. Και θα μάθουμε, τότε θα μπορέσουμε να δούμε ποιους στόχους καλούμεθα να εκπληρώσουμε. Και αν πετύχουμε να το κάνουμε, τότε θα προωθήσουμε αυτή τη συζήτηση που το ή άλλως βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεύτερη παρατήρηση. Κοιτάξτε ακριβώς το κείμενο το οποίο εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ το κοίταξα και έχω την εντύπωση ότι οι πολιτικές ομάδες συμπεριέλαβαν κάποιες παραγράφους για το Δούναβι που νομίζω ότι χαράσουν μια κατεύθυνση. Ε, μπορεί κανείς να διερωτηθεί για το ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι, αλλά νομίζω ότι οι παράγραφοι αυτοί μπορούν να μας ε, βοηθήσουν και με τώρα από αυτά μπορούμε να διευρύνουμε και την οπτική μας γωνία. Ίσως ε, το διατύπωσα κάπως γενικά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και τον κύριο Κούν από την Επιτροπή Μεταφορών, γιατί η Επιτροπή Μεταφορών συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία ε, προετοιμασίας γνωμοδότησης. Τον παρακαλώ λοιπόν να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκε ότι σήμερα συζητούμε για αυτό το θέμα, μπορούμε να συζητήσουμε μάλλον για αυτό το θέμα, επειδή η Σουηδική Προεδρία τότε ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία από κοινού με την αρμόδια επίτροπο, την κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ, που τώρα είναι πρόεδρος αυτής της επιτροπής. Και πραγματικά έκανε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και ε, πράγματι τα πράγματα θα πρέπει να πάνε προς τα εκεί, ώστε να έχουμε ένα πρόγραμμα υπόδειγμα. Ε, ευχαριστούμε για την ε, έκθεση του κυρίου Ολενίτσακ. Ε, μπορεί να μας ασμεύσει σαν βάση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συγκεντρωθούμε στις ε, μεγαλύτερες προτεραιότητες όσον αφορά τη Βαλτική που καταρχήν είναι το περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερος ευαίσθητο θέμα. Θα πρέπει να υπάρξει μια οικολογική ισορροπία στη Βαλτική. Γιατί είναι οι πηγές μας, οι πόροι μας. Αν σκεφτούμε την αλία ή τον τουρισμό, τι γίνεται εδώ. Ε, έγινε λόγος για τις πλωτές ε, μεταφορές. Θα πρέπει να δούμε όμως, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με το περιβάλλον. Γιατί Εάν μιλάμε για οικονομία για τις γειτονικές χώρες, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα αστικοποίησης, υπάρχουν απόβλητα των βιομηχανιών κλπ. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα υποστηρίξουμε με τις απαιτούμενε επενδύσεις στις υποδομές. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, ευημερία, επίσης ζήτημα κεντρικής ε, σημασίας. Και η ευημερία σχετίζεται με το πώς μπορούν οι άνθρωποι στην περιοχή της Βαλτικής να ζουν ευτυχείς και να έχουν και επαρκή εισοδήματα. Όλα αυτά σχετίζονται με θέματα της οικονομίας. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ε, ποιους ε, πυρήνες της οικονομίας θέλουμε να προωθήσουμε στη Βαλτική. Βεβαίως η ναυτική οικονομία έχει μεγάλη σημασία, αλλά και οι κατασκευές, γιατί είμαστε στην ευτυχή θέση και εγώ είμαι μηχανικός, να έχουμε ε, θέσεις εργασίας ε, στον τομέα των κατασκευών ή, της ναυπηγ... τα ναυπηγεία. Ε, υπάρχουν έτοιμε θέσει εργασία. Χρειαζόμαστε γερανού για τη μεταφορά των πλοίων κλπ. Τώρα, το πώς θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Αυτά συνδέονται με, τους, με τα συγκοινωνιακά δίκτυα το σημείο λοιπόν αυτό είναι τέλος καθοριστικό. Θα πρέπει λοιπόν στα δική να συμπεριλάβουμε του επενδυτικού πόρους για τη βελτίωση των διευρωπαϊκών δικτύων, για τον τομέα μεταφορά για το δικό δίκτυο, για τους σιδηροδρόμους, αλλά και για τις ε, πλωτέ συγκοινωνίε. Και για τον τουρισμό επίσης το ζήτημα της ε, συμφόρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ένας τουρίστας που έρχεται σε αυτή την περιοχή και εγκλωβίζεται στη συγκοινωνία, ε, εγκλωβίζεται στο δρόμο, δεν θα πρόκειται να το επαναλάβει λόγω κυκλοφορικής συμφόρησης, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναεπισκεφθεί αυτή την περιοχή. Τώρα, το σημείο της ασφάλειας. Η ασφάλεια παίζει από την έννοια αυτή κεντρικό ρόλο. Εάν δούμε ποια είναι η κίνηση των πλοίων σε αυτή την ε, θάλασσα που είναι η θάλασσα με το πιο πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών, η Βαλτική. Εδώ ε, είχαμε ήδη και στο παρελθόν δυσκολίες. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία όσον αφορά τη μεταφορά του αργού πετρελαίου ε, έχει κατά νου τη Βαλτική. Εγώ, η πατρίδα μου είναι η Πομερανία. Εκεί γεννήθηκα στην νότια ακτή της ε, Βαλτικής, 400 μέτρα από τη θάλασσα και γνωρίζω. Εκεί θα πρέπει να έχουμε μια, να εγκαταστήσουμε ραντάρ για να δούμε τι γίνεται με τα ατυχήματα των ε, τάνκερ και τις ε, πετρελοκυλίδες από τα ρώσικα φορτηγά, για παράδειγμα, που ρηπαίνουν τη Βαλτική. Αυτό σχετίζεται και με ζητήματα του τουρισμού. Αυτή είναι η συγκεκριμένη παρατήρηση που ήθελα να κάνω. Ε, τα, οι συγκοινωνικές οδοί ε, μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων ε, συνδέονται με τα σημεία διανομής του εμπορίου μέσω των λιμένων. Αυτά είναι τα σημεία διασύνδεσης ε, μέσω της Βαλτικής. Μπορεί να φτιάξει κανείς ε, μεγάλες γέφυρες, αλλά μπορεί με τις πλωτές συγκοινωνίες, ε, με τις πλωτές μεταφορές να έχει εξαιρετικά δίκτυα διανομή. Η δική μου πρόταση είναι από αυτή ακριβώς την οπτική γωνία και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όσον αφορά την Περιφερειακή Επιτροπή και τα ερωτικά τομεία να φτιάξουμε ένα μοντέλο χρηματοδότησης, γιατί μόνο με ένα ή δύο εκατομμύρια δεν θα τα καταφέρουμε, όπως είπε και ο κύριος Όλμπριχτ και ο κύριος Ολενίτσακ επίσης. Θα πρέπει από κοινού να προβληματιστούμε για το ότι χρειαζόμαστε κονδύλια, χρειαζόμαστε ένα προπολογισμό για την ανάπτυξη της Βαλτικής. Μπορούμε να βρούμε αυτά τα χρήματα από διάφορες ε, πηγές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε να κάνουμε τη Βαλτική υποδειγματική περιοχή. Και αν η περιοχή του Δούναβη και η περιοχή της Μεσογείου ε, ε, προσελκύσουν επίσης το ενδιαφέρον μας, φέρουμε εδώ πολύ μεγάλη ευθύνη. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο δεν γνωρίζουμε ε, τέτοια ζητήματα χωροταξίας όπως έχουμε σε εθνικό επίπεδο αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε αυτές τις πτυχές ε, ε, χωροτακτικής πολιτικής. Για παράδειγμα, όσον αφορά την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου οι ε, αγωγούς ε, ηλεκτρικού ρεύματος. Ε, να δούμε πού θα πρέπει να εγκατασταθούν μακριά, από την ακτή και λοιπά ή σε πιο ακριβώς σημείο. Να δούμε ποιες θα είναι οι ενδεδειγμένες περιοχές για τον τουρισμό, ποιες είναι οι περιοχές που ανδείκνονται για την αλία ε, και ποιες είναι οι οικολογικά ευαίσθητες περιοχές που θα πρέπει να προστατεύονται. Ε, κάτι τέτοιο γίνεται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το δίκαιο. Ε, ίσως θα πρέπει να το κάνουμε και για την Βαλτική. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής πριν πάρει το λόγο η Επιτροπή Thank you very Είναι ο κύριος Γκοντμάνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2008 ε, έγινε το Συμβούλιο της ε, Βαλτικής, όταν εμεί είχαμε την ε, Προεδρία και συζήτησαμε τα θέματα αυτά και ο κύριος Μπαρόζο συμμετείχε και υπήρχαν σημαντικά θέματα ενέργειας, επίσης τα ζητήματα ενός αγωγού φυσικής, ε, φυσικού αερίου κλπ. Επίσης ήμουν σε συνεδρία του Συμβουλίου όταν τέθηκε το θέμα για την ε, Μεσογειακή Ένωση, για την Ένωση της Μεσογείου. Ε, Βεβαίω αυτά είναι δύο εντελώ διαφορετικά θέματα, όσο παρόλα αυτά παρουσιάζουν ορισμένε ομοιότητε η περιοχή της ε, Βαλτικής και η Μεσόγειας έχουν μια, μια, ένα κοινό σημείο όσον αφορά τη σχέση με τις γειτονικές ε, χώρες και είναι σημαντικό να διορθωθούν οι σχέσεις με τις χώρες που βρίσκονται νοτίως της Μεσογείου και βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για την στρατηγική της Βαλτικής ε, σε σχέση με χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόβλημα υπαρθμών ένα που ανακύπτει είναι ακριβώς η χάραξη μιας πολιτικής γειτονίας. Ε, νομίζω ότι ε, δεν έγιναν πολλά πράγματα. Ε, λέχθηκαν πολλά πράγματα, αλλά δεν κατέστη σαφές πώς θα προβούμε στην εφαρμογή. Και για να είμαστε έντιμοι, είναι επικίνδυνα θέματα. Γιατί αν αυτές οι μακροπεριφέρειες αν, υπάρχει μια εφαρμογή σε σχέση με τις μακροπεριφέρειες, θα υπάρξει ένας φθόνος από οικονομική άποψη, ε, γιατί οι περιφέρειες αυτές θα αναπτυχθούν πολύ γρήγορα, η Βαλτική, ο Δούναβης κλπ. Και το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την πολιτική συνοχή και τη χρηματοδότηση αυτών των πραγμάτων. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινεί, λοιπόν. Στα διευθυντικά ταμεία έχουμε μια γραμμή που λέγεται ε, γραμμή προπολογισμού για πολλές ε, χώρες και που χρηματοδοτείται από Ταμείο Συνοχής. Πρόκειται για προγράμματα που αφορούν πολλές χώρες. Ε, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες βέβαια γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών. Και όταν μιλάμε για τέτοιες περιφέρειες, δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερα πολλά έκτακτα κονδύλια. Συνεπώς, αν μιλάμε για τη Βαλτική, η Βαλτική θα υπαχθεί σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού που αφορά ταυτοχρόνως πολλές χώρες. Και αν μιλάμε για άλλες χώρες, για την, ε, ε, για την ε, χάραξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχουν κάποια προγράμματα Interreg, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί οι χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι ιδιαίτερως ευτυχείς για την δαπάνη αυτών των χρυπάνων. Και νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αφορούν τις μακροπεριφέρειες. Οι λόγοι αυτοί διαφέρουν για τις διάφορες περιοχές. Ε, ε, στη Βαλτική έχουμε μεγάλη μόλυνση. Ε, ακόμα και το ΝΑΤΟ έκανε μια ανάλυση για το ποιο θα ήταν, πόσο υψηλό θα ήταν το κόστος του καθαρισμού των υδάτων της Βαλτικής και είναι εξαιρετικά υψηλό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Υπάρχουν ε, άλλες χώρες που, υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν είναι πολύ ανεπτυγμένες και θα ήταν ιδιαίτερως ευτυχεί να δεχθούν κάποια οικονομική βοήθεια. Επίσης υπάρχει το θέμα των σχέσεων με τις γειτονικέ χώρες. Εγώ είμαι ιδιαίτερο συντηρητικός όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα οικονομικής αποκέντρωσης που θα οδηγήσει σε φαινόμενα φθόνου. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εμείνουμε στις βασικές κατευθυντήριες ε, γραμμές του Ταμείου Συνοχής και θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να συμπεριληφθούν στη γραμμή προϋπολογισμού που αφορά πολλές χώρες ταυτοχρόνως. Δεν θα δημιουργηθεί άλλη γραμμή προϋπολογισμού. Δεν είμαι υπέρ του να δημιουργηθεί άλλη γραμμή προϋπολογισμού. Ε, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον προπολογισμό του 2010, πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Εάν τα χρήματα αυτά χρησιμοποιηθούν μόνο από ορισμένε χώρε, να τα πάρουν και να τα χρησιμοποιήσουν με ένα οποιοδήποτε τρόπο, νομίζω ότι οι άλλε χώρε δεν θα είναι ιδιαίτερα ευτυχεί αν συμβεί κάτι τέτοιο. Συνεπώ λοιπόν τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα και εγώ το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Γιατί έγινε για παράδειγμα προτάσει να υπάρξουν αποκεντρωμένε σχέσει με τι χώρε τη Ανατολική ε, Μεσογείου, τη Ενωτίου Μεσογείου, συγγνώμη. Ε, Νοτιοανατολικής ε, Μεσογείου. Ε, ε, εδώ υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι. Νομίζω ότι δεν έχουμε ένα καινούριο μοντέλο. Εγώ είμαι τελείως ξεκάθαρο. δεν θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον γραμμή στον προπολογισμό, αλλά θα πρέπει να υπαχθεί στην υπάρχουσα γραμμή του προπολογισμού και θα πρέπει να παραμείνουμε στο υφιστάμενο ε, σύστημα μέχρι το 2013 εκτός εάν δημιουργήσουμε ένα νέο σκεπτικό και κάποιο μηχανισμό ικανό να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Εάν δεν το πράξουμε θα έχουμε σοβαρά προβλήματα νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί και συντηρητικοί στο σημείο αυτό. Εάν δεν το κάνουμε θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Ο David Sweet από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως ο Δαβίδ θα ήθελε να διευκρινίσει λιγάκι καλύτερα τα θέματα αυτά μετά από τις ερωτήσεις των συναδέλφων, ιδίως σε σχέση με το ζήτημα της χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά πάντα να έρχομαι ενώπιον τη Επιτροπή σα για να μιλήσουμε για τι περιφερειακέ στρατηγικέ. Όχι μόνο επειδή μα αρέσει να μιλάμε για το έργο μα, γιατί βρισκόμαστε στο κατάλληλο σημείο εκεί που υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη για τα θέματα αυτά. Δεν χρειάζεται να σα εξηγήσω τι βασικέ αρχέ ή οτιδήποτε τέτοιο. Νομίζω ότι η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο η πολιτική υποστήριξη, το να πείτε ότι είναι θετικά όλα αυτά, αλλά και οι συγκεκριμένε οι πρακτικέ προτάσει, ε, οι προτάσει για λύση που έρχονται από εσά είναι πάρα πολύ σημαντικέ και χαιρόμαστε για όλα αυτά τα θέματα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να καθησυχάσω αυτού από εσά που νομίζετε ότι δεν έχει γίνει τίποτα από το περασμένο καλοκαίρι με τι παρουσιάσει και τι συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συνάντηση στη Στοκόλμη, όπου ήμουν παρόν εγώ, με την παρουσία των εθνικών σημείων επαφή από τι χώρε τη περιοχή τις οκτώ χώρες που ήταν ε, παρούσες και επίσης με τους συντονιστές από τα 15 <clears throat> κέντρα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Εξετάσαμε θέματα προτεραιότητας, είδαμε αν προχωρούν τα σχέδια, αν υπάρχουν σημεία συμφόρησης, αν υπάρχουν ε, προβλήματα να εντοπίσουμε τον κατάλληλο συνομιλητή σε ένα κράτος μέλος ή αν δεν υπήρχε κατάλληλη χρηματοδότηση. Ο στόχος ήταν να βρούμε, να εντοπίσουμε ποιος θα έπρεπε να αναλάβει την λύση των προβλημάτων του κάθε προβλήματος και να βρούμε τους συγκεκριμένους τρόπους να προχωρήσουμε από τη σκέψη στη δράση και να εξασφαλίσουμε ότι τα σχέδια αυτά θα γινόταν πραγματικότητα. Η εμπειρία μου δείχνει ότι είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει ο συνδυασμός μιας εθνικής δράσης εκ των άνω προς τα κάτω με συμμετοχή σημείων επαφής που λειτουργούν σε ένα πιο βασικό επίπεδο. Όλοι αυτοί να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά από κοινού. Όλοι θέλουν να έχουν χρηματοδότηση, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός η χρηματοδότηση, γιατί και αυτό είναι τμήμα της, ε, των υπολογισμών, της αριθμητικής, αν θέλετε, της στρατηγικής της Βατικής. Ανακαλύψαμε ότι οι λύσεις πρέπει να βρεθούν μέσα στους διαθέσιμους πόρους για την περιοχή αυτή. Γι' αυτό είπαμε όχι νέα χρήματα, αλλά συγχρόνως και όχι νέοι φορείς και όχι νέα νομοθεσία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες δομές, νέες γραμματείες, νέους φορείς κτλ. Απλώς να συνενώσουμε τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στην περιοχή. Πού βρισκόμαστε λοιπόν μετά από όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι η Κομισιόν εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική δεν θέλουμε να διευρύνουμε με μεγάλη ταχύτητα όλα αυτά τα θέματα και να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη μακροπεριφερειών, εκτό αν είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι ο καλύτερο δρόμο προ τα έμπρο. Ορισμένοι από εμά είμαστε πεπισμένοι. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δούμε θετικά αποτελέσματα από το παράδειγμα τη Βαλτική και τι άλλε υποανάπτυξη μακροπεριφέρειε. Πολλοί από εσά έκαναν σαφές ότι μπορεί να προκύψουν δυσκολίες αν υπερεπεκτείνουμε την πορεία αυτή των μακροπεριφερειών. Παραδείγματος χάρη, είναι φανερές οι δυσκολίες που έχουμε αν θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή την έννοια σε περιοχές όπως η Μεσόγειος. Δεν θέλουμε λοιπόν να τρέξουμε πρωτού μπορούμε να περπατήσουμε, ούτε να θέσουμε το άρωτρο πριν από το βόδι. Αυτό το οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι να έχουμε κάτι το οποίο είναι λειτουργικό και μετά μπορούμε να δούμε αν αυτό το παράδειγμα μπορεί να μεταλαμβαδευτεί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Και γι' αυτό θέλω να μπω τώρα σε θέματα λεπτομεριακά προϋπολογισμού και στρατηγικής που θα έχουν σημασία για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές. <clears throat> θέλω όμως να τονίσω ότι έχω απόλυτη κατανόηση για αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να είναι χρήματα τα οποία θα κατανεμηθούν στα κράτη-μέλη με βάση προράτα, βάση σαφών σαφώς καθορισμένων κανόνων. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν λεπτομεριακές γεωγραφικές ε, διαρρυθμίσεις και κανόνες ε, επιλεξιμότητος. Θα ήταν πρόσφορο λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση. Τέλος, για τα 20 εκατομμύρια τα οποία ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό του 2010, η Κομισιόν εξετάζει ακόμα με πιο καλύτερο τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα και αυτό δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο, γιατί να μην χαιρόμαστε απλώς που μας δίνετε αυτά τα λεφτά. Γιατί αν έχετε εκατομμύρια, <clears throat> ακόμα και 20 εκατομμύρια, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο για την εκταμείευση αυτών των ε, ποσών. Να υπάρχει ένα δίκαιο και ανοιχτό και σαφές πλαίσιο που θα εξασφαλίσει ότι ακόμα και για τα πιλωτικά προγράμματα ότι υπάρχει μια σωστή σχέση κόστους-οφέλειας. Και δεν είμαστε σίγουροι ότι ακόμα μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τους τωρινούς κανόνες του προϋπολογισμού. Δεν θα σας κουράσω με αυτά τα θέματα τα οποία τα γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε τώρα να ενισχύσουμε ενδεχομένω το υπάρχον διακρατικό διασυνοριακό πρόγραμμα για την αυτιλία στην Βαλτική ή να ενισχύσουμε το πρόγραμμα για τη βόρεια διάσταση όπου εμπλέκεται και η Ρωσία. Σε 10 μέρες θα πάμε στη Ρωσία για να δούμε σε υψηλό επίπεδο ποια είναι τα προβλήματα που είναι οι φραγμοί και πώς μπορούμε να τους ξεπεράσουμε ώστε να υπάρξει καλύτερη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Χρειαστήκαμε πολύ χρόνο, αλλά προχωρούμε προς την κατεύθυνση αυτή και ξέρουμε πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και ξέρουμε ότι δεν θα είναι επιτυχής αυτή η στρατηγική, εκτός αν μπορέσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν και άλλε δυνατότητε να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα καλύτερα χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία θα λειτουργήσουν ως καταπιστευματίες για αυτά τα χρήματα και στη συνέχεια μπορούν να δοθούν για σχέδια που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλες πτυχές, από άλλες πλευρές μάλλον. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά. Έχουμε φυσικά το πρόβλημα του χρονοδιαγράμματος του προϋπολογισμού και να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε πόσα μέχρι μια καταληκτική ημερομηνία. Δεν ξέρω λοιπόν ποια δομή θα πάρει αυτή η χρηματοδότηση, τα εξετάσουμε όλα αυτά, αλλά ο στόχος μας είναι να έχουμε μία λύση που δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βολέψουμε αυτά τα 20 εκατομμύρια τα οποία δεν περιμέναμε και να τα κατανείμουμε σε όλους, αλλά να είναι μία πραγματική οδός που μπορεί να ακολουθηθεί όταν οι αρχές του προϋπολογισμού θεωρήσουν ότι πράγματι αξίζει να προχωρήσουμε. Σας έχω επεκταθεί ίσω πολύ, αλλά τονίζω και πάλι ότι είναι μεγάλη χαρά για μα να μπορούμε να συζητούμε αυτά τα θέματα είτε σε διμερή επίπεδο είτε ενώπιον μια επιτροπή όπω η δική σα. Ευχαριστούμε πολύ, Ντέβιτ. Πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση τώρα αυτή. Θα έχουμε τη συζήτηση για το σχέδιο έκθεση στην κανονική μα συνεδρίαση του Μαρτίου. Αν κυρία Ολενίτσο εκθέτουν να κάνετε τώρα κάποιο σχόλιο, ευχαρίστω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει προτάσεις, έχουν διατυπώσει σχόλια. Από τη δική μου πλευρά θέλω να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι αυτή η πολιτική απαιτεί συνεργασία για τις μακροπεριφέρειες, απαιτεί κοινό καθορισμό στόχων για τις μακροπεριφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από την ε, συγκεκριμένη αυτή περιοχή που θέλουμε να καλύψουμε και την εμβέλεια των μέτρων και επίσης σε σχέση και με τις δυνατότητες του προπολογισμού. Αυτές οι ανάγκες <clears throat> θα πρέπει να δούμε πώς θα καλυφθούν. Μπορούν να καλυφθούν από εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο και με μία στοχοθεσία που θα εξασφαλίσει κάποιες προτεραιότητες για, τους, για τα κονδύλια αυτά, τα οποία θα δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη-μέλη αυτά. Επίσης, θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητες αυτά τα θέματα των μακροπεριφερειών, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, τι θα γίνει με τη διαδικασία συγχρηματοδότησης σε επίπεδο μακροπεριφερειών. Θα είναι ένας πρόσθετος ε, προϋπολογισμός, ένας διευρυνθμένος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να διαλευκανθούν σε ένα μέλλον όχι κατά ανάγκη άμεσο μέλλον, αλλά σε ένα ορατό μέλλον. Και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν μέσα σε μια κοινή προσπάθεια εξέβρεσης εξωτερικών κονδυλίων από την Παγκόσμια Τράπεζα, πράγματος χάρη, ή από επενδύσεις άλλων χρηματοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο σύνολο των ερωτηματών αυτών για να καθορίσουμε ποια ακριβώς θα πρέπει να είναι η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτό το κοινό εγχείρημα. Και πρέπει να είναι κοινό εγχείρημα γιατί η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πια μια πραγματικότητα και θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινέ προκλήσεις, αυτά τα κοινά καθήκοντα, ιδίως όταν ξεπερνούν τα τωρινά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Ολενίτσεκ. Πιστεύω ότι το Μάρτιο θα αντιμετωπίσουμε πράγματι αυτή την προ... πρόκληση να είμαστε συγκεκριμένοι στην γνωμοδότησή μας για το πώς βλέπουμε την στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βαλτική και γενικά για τις μακροπεριφέρειες. Ξέρουμε ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος επίτροπος το Φεβρουάριο κατά ψευθανότητα και μπορούμε να αναμείνουμε την πρόταση της Κομισιόν και μετά να αντιδράσουμε ή όπως προτείνεται μπορούμε ήδη στην έκθεση του κυρίου Ολενίτσεκ να συμπεριλάβουμε κάποιες δικές μας προτάσεις. Απλώς σας λέω ότι έχουμε δύο επιλογές. Ή θα πούμε, ή θα πρέπει να πούμε ότι τέτοιου είδους μακροπεριφερειακές πολιτικές μπορούν να γίνουν και επίσημα τμήμα του τρίτου στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν στο παρελθόν το Interreg, να γίνει τμήμα λοιπόν της ε, διαμεθοριακής πτυχής αυτής της πολιτικής. Και φυσικά αυτά θα πρέπει να καθοριστούν μέσα σε διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη και να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω. Μάλλον έχει ακολουθηθεί μια διαδικασία εκ των άνω προς τα κάτω. Εμείς θα θέλαμε να ενισχύσουμε τη διαδικασία εκ των κάτω προς τα άνω, να προσκαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλευτεί περισσότερο με τις ε, περιφέρειες για να δούμε ποια είναι τα αναδυόμενα κοινά προβλήματα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι τμήμα της διαμεθοριακής αυτής συνεργασίας μέσα στην πολιτική ε, συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα πλαίσιο για να δώσουμε τη δυνατότητα στα, στις περιοφέρειες αυτές που θέλουν να έχουν μια βαθύτερη διασυνοριακή συνεργασία να το πράξουν. Και ίσως υπάρχουν και άλλες επιλογές τις οποίες θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη. Πάντως θα πρέπει το Μάρτιο να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε με τις συστάσεις μας και ενδιαμέσως θέλω να σας πω ότι προσεκλήθηκε εγώ στο Ούλμα στις 2 Φεβρουαρίου όπου λαμβάνει η χώρα μια συνάντηση επίπεδου με συμμετοχή επιτρόπων για την Δουνάβια στρατηγική και θα είμαι παρούσα στην τελική σύνοδο τη συνδιάσκεψη αυτή. Επομένω, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη προχωρούν και συμμετέχουμε όλο και περισσότερο στο επόμενο εγχείρημα που είναι η στρατηγική του Δούναβη. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Όλα και Θα συζητήσουμε περαιτέρω για το θέμα αυτό το Μάρτιο και νομίζω ότι έχετε προσκαλέσει τους αδέλφους άτυπα να συζητήσουν μαζί σας κύριε Ολανίτσεκ. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πρωτού προετοιμάστε το τελικό του έγγραφο. Τελευταίο σημείο της ημέρας διάταξης. Ο κύριος Λαμπέρφαν Νίστλεροι ανταλλαγή απόψεων για την έκθεσή σας σε σχέση με τις συνέργειες μεταξύ της ε, περιφερειακής και της ε, πολιτικής συνοχής και κύριε Φανίς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να κάνουμε ε, συζήτηση για δεύτερη φορά ε, επί του εγγράφου εργασία. Απλώ να σα δώσω κάποιε πληροφορίε όσον αφορά τι ε, πρόοδου που έχουμε κάνει. σχετικά με την έκθεση αυτή. Και όπως γνωρίζετε, Πρόκειται και για τον ε, κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες. Ε, μιλάμε εδώ για υλοποίηση ε, υφισταμένου προγράμματος με στρατηγικές που πρέπει να αναπτυχθούν αλλά παρόλα αυτά το νομικό υπόβαθρο είναι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς θα γίνει η υλοποίηση και εάν ε, μπορούμε να κάνουμε κάποιες ε, συστάσεις ε, και για τα δύο σημεία. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθαμε σε επαφή με τους συναδέλφους της Επιτροπής Ήτρε η οποία Επιτροπή έχει πλήρη αρμοδιότητα όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη κυρίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό έπρεπε να δούμε πώς θα, γίνει η συνεργασία μας, πώς θα μπορούμε να ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες μας. Και τελικά συμφωνήσαμε μετά από μια σειρά καλών διαπραγματεύσεων να ε, εφαρμόσουμε τον ε, κανονισμό 50 του ιστορικού κανονισμού για την ε, Ήτρε, του, του κανονισμού the one committee and one of the others and διαδικασίας για την Ήτρε. Και μπορώ να πω ότι οι περιφέρειες Ρέτζι και Ήτρε έχουν συμφωνήσει για τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τους κανονισμούς και αναγνωρίζοντας τους στόχους ε, της πολιτικής έρευνας και συνοχής ε, και αποφάσισαν ότι θα πρέπει να ε, έχουν ισότιμη θέση. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ασχολείται περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις συνεργίες ανάμεσα ε, στις, στα ε, ταμεία και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα ε, και την ανάπτυξη, καθώς επίσης και με τα προγράμματα καινοτομίας και ανάπτυξης. Τώρα, η Επιτροπή ΙΡΤΡΕ θα έχει άλλες αρμοδιότητες, δηλαδή θα αναλύσει τις, ε, τα προγράμματα και τις στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης και θα έχουν και κοινέ δραστηριότητες, δηλαδή θα αναλύουν και θα κάνουν συστάσεις ε, σχετικά με τον συντονισμό ανάμεσα ε, στην πολιτική συνοχή και την πολιτική έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι η Ήτρε βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο κατά κάποιο τρόπο ε, με την Επιτροπή Ρέτζη. Έχει ορίσει τον κύριο Χατζημαρκάκη ως ε, εισηγητή και συμφωνήσαμε επί της διαδικασίας, πράγμα που σημαίνει ότι ε, το δικό μου προσχέδιο ε, θα υποβληθεί προς εξέταση τον Μάρτιο στην, Επιτροπή, ε, της, στην συνάντηση της Επιτροπής μας και θα ψηφιστεί 26-27 ε, Απριλίου. Όσον αφορά τώρα την Επιτροπή Ήτρε, το προσχέδιο θα εξεταστεί τον Φεβρουάριο και στις 17-18 Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί. Επομένως, ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες όσον αφορά όχι το περιεχόμενο της έκθεσής μου, αλλά όσον αφορά τη διαδικασία. Γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό και εργαζόμενοι δηλαδή ε, και στις δύο επιτροπές, Ήτρε και ε, Ρέτζι, ε, θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη τοποθέτηση απέναντι στα εργαλεία συνοχής καθώς επίσης ε, και όσον αφορά τα εργαλεία του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτά ήταν διαδικαστικά τα ζητήματα και ε, νομίζω ότι αν λειτουργήσει ε, το σύστημα θα είναι πάρα πολύ καλό γιατί διαφορετικά εμείς θα λέμε είμαστε η Επιτροπή Ρέτζη και είμαστε οι πρώτη και οι καλύτεροι ενώ η Επιτροπή Ήτρα θα λέει ε, αντίστοιχα τα ίδια. Επομένως τώρα καταφέραμε να καταμερίσουμε τις αρμοδιότητες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν μια κοινή βάση, μια κοινή πολιτική βάση για το μέλλον. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα, εάν θέλετε τώρα τι γίνεται ακριβώς, τι προβλέπει ακριβώς ο κανόνας 50 ε, και τα λοιπά, νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω ένα γραπτό υπόμνημα τις επόμενες μέρες. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστούμε. Ένας ε, ο αγορητής έχει εγγραφεί, δεν ξέρω αν θέλουν και κάποιοι άλλοι. Παρακαλώ. Um, ναι, Λαμπέρτ, Δύσκολο είναι αυτό να καταλάβει κανείς τι βρίσκεται πίσω από αυτό τον τίτλο. Εγώ τι θα ήθελα. Να σκεφτούμε περισσότερο ποιο θα έπρεπε να, να είναι αυτό που θα κάνει το πρόγραμμα πλαίσιο για να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στην πολιτική συνοχή. Δεν θα ήθελα να το αφήσω αυτό στους συναδέλφους μας της Ήτρε. Αυτό είναι δική μας αρμοδιότητα, δικό μας αγροτεμάχιο. Αλλά αν κοιτάξουμε τον τίτλο τον οποίο έχουμε ενώπιόν μας και τον πίνακα μάλλον, να δούμε αν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι και τα θέματα της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα αυτά είναι δική μας αρμοδιότητα. Δεν συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με αυτά που είπες Λαμπέρ. Εντάξει, καλά. Το επόμενο το ερώτημα είναι τι θέλουμε να αποκομίσουμε από αυτήν την έκθεση. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό εν ώψη της επόμενης περίοδου προγραμματισμού μετά το 2013. Εγώ θα ήθελα ένα σημαντικό τμήμα της εργασίας μας για την έκθεση αυτή είναι να εξετάσουμε το θέμα του προσδιορισμού, του earmarking. Είναι αυτή η καλύτερη μέθοδος για το μέλλον. Και δεύτερον, ποια είναι η στοχοθεσία που ακολουθούμε. Τι είδος έρευνας, τι είδος στρατηγικής θέλουμε. Πώς συνδέεται αυτό με την Ευρώπη 2020. Και τι σημαίνει αυτό και ό,τι αφορά τη στρατηγική έρευνας. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Γιατί τα προγράμματα πλαίσια, τα, το, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα έχει κάνει κάποιες ε, μελέτες οι οποίες κοιτάζουν πώς θα αντιμετωπιστεί και θα συνεχίσει η εκμετάλλευση του άνθρακα, κάτι το οποίο μπορεί να μην ευνοεί συγκεκριμένα τις περιοχές αυτές που έχουμε ενώπιον μας. Αν θέλουμε να έχουμε μια αηφόρο ανάπτυξη στις περιοχές αυτές δεν πρέπει να δούμε με αυτούς τους στόχους την έρευνα. Αυτό εννοώ όταν μιλάω για τη στοχοθεσία και το τελευταίο ζήτημα έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση. Θα χρηματοδοτήσουμε όλες τις ερευνητικές ενέργειες ή μονάχα τις ενέργειες, τις έρευνες οι οποίες είναι μελλοντόστροφες και επίσης ποιες θα είναι και οι συμβολές της περιφερειακής πολιτικής για τα κέντρα αριστείας. Και εξάλλου, πού θα βρεθεί το προσωπικό για τα κέντρα αριστείας. Ποια είναι η προϋπόθεση για να έχουμε άνθρωπους, προσωπικό, ερευνητές που θα στελεχώσουν τα, τα κέντρα αυτά αριστείας. Πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτό το θέμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει στο έγγραφο εργασίας σου. Θα ήταν πολύ καλό να προσθεθεί και αυτή η προβληματική λοιπόν Και κατά τα άλλα είπαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την οικολογική και την οικονομική και την κοινωνική πτυχή. Να έχουμε περιφέρειες με κέντρα αριστείας λοιπόν που θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ε, Ήθελα μια σύντομη παρουσίαση, μια σύντομη μάλλον ένα σύντομο σχόλιο στο, στα όσα υπόθηκαν εισαγωγικά και στην έκθεση που έχουμε μπροστά μας. Ε, προσωπικά νομίζω ότι δεν είναι σαφές τι ακριβώς αποσκοπούμε. Έχω τη γνώμη ότι δημιουργία κέντρων αριστείας έρευνας στην περιφέρεια και αξιοποίηση ε, κοινοτικών κονδυλίων για αυτή την κατεύθυνση ή ακόμα και των ερευνητικών προγραμμάτων δεν οδηγεί πάντα και κατά ανάγκη σε σύγκληση της περιφέρειας. Τουλάχιστον τα κριτήρια που έχουμε θεσπίσει μέχρι τώρα. Ε, το κριτήριο που θα οδηγούσε στη σύγκριση θα ήταν κατά τη γνώμη μου η σύνδεση μιας περιφερειακής έρευνας, μιας έρευνας που γίνεται στην περιφέρεια με μια παραγωγή στην περιφέρεια. Εκεί ναι, μπορεί να ελπίζει κανείς ότι σιγά σιγά η έρευνα θα συμβάλλει στον να το επίπεδο της ε, περιφέρειας. Ε, βλέποντας όμως ε, το κείμενο της έκθεσης και ιδιαίτερα στη σελίδα 4 που γίνεται λόγος ότι σκοπός είναι ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι να οθήσουμε τις περιφέρειες σε έναν ανταγωνισμό ποιες από αυτές θα δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες για κέντρα ε, αριστείας στην έρευνα. Και αυτό, επαναλαμβάνω, και από μια πρακτική που υπάρχει ήδη, είναι γνωστά ορισμένα παραδείγματα, ειδικά σε αναπτυγμένε χώρε τη Δυτική Ευρώπη, αλλά και από αλλού δεν θα οδηγήσει κατά ανάγκη στην ε, σύγκληση και στην ανάπτυξη τη ε, περιφέρειας. Ε, νομίζω αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαριστούν, ε, διότι διαφορετικά και η Επιτροπή Αρμόδια για την Έρευνα και Τεχνολογία θα νομίζει ότι πάμε να πάρουμε χρήματα <laughs> από τα δικά του προγράμματα και εμεί δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα ε, γιατί προφανώς είναι σκοπός αυτός. Και ένα δεύτερο, ε, προφανώς ε, τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία μας απασχολούν πρέπει να ανταποκρίνονται σε ανάγκες των περιφερειών, σε ανάγκες των εργαζομένων, στις ανάγκες των αγροτών και σε διάφορα άλλα που πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν στο γενικό πρόγραμμα πλαίσιο της ε, κοινότητας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you. Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στόιρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι την... δεν συμμερίζομαι την κριτική της κυρίας Σρόντερ. Έχω ρητά την άποψη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα στο ζήτημα έρευνα και καινοτομία. με τους συναδέλφους στην Ήτρε να συζητηθεί. Το, βέβαια το ερώτημα είναι ποια θα είναι η έκβαση αυτών των συζητήσεων. Αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Αλλά ωστόσο, εάν εγερθεί το θέμα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και με την Ήτρε. Ο κύριος Χάν, ο κύριος Επίτροπος στην Ακρόαση εξέφρασε μια, απόφαση, μια άποψη η οποία θεωρώ ότι αξίζει να την σκεφτούμε. Είπε ότι η έρευνα της αριστείας δεν, μπο, δεν χρειάζεται να περιοριστεί σε έναν τόπο, αλλά μπορεί να γίνει παντού στην Ευρώπη. Βεβαίω, η προσέγγιση τη περιφερειακής πολιτική είναι διαφορετική, γιατί εμείς λέμε ότι θέλουμε να υπάρχουν ε, σε ορισμένε περιοχές, σε ορισμένοι θεσμοί. Ε, Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη τι συνέργειε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κοινή προσέγγιση αλλά από την άλλη θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα σημεία τομή ή που είναι οι διαφορέ μια ερευνητική στρατηγική που πηγαίνει στην κατεύθυνση αριστείας και μια στρατηγική που εξυπηρετεί του στόχου τη περιφερειακή πολιτική, δηλαδή την αποκέντρωση. Και εδώ σκέφτομαι ότι έρχεται η καινοτομία στο επίκεντρο, γιατί όπω κατάλαβα εγώ τα πράγματα, οι λιγότερε καινοτομίε και οι λιγότερες ε, ανακαλύψεις βάσης που αφορούν τεχνολογία βάσης ε, δεν ε, δημιουργήθηκαν μέσω μιας συγκεντρωτικής προσέγγισης αλλά αντίθετα αποκεντρωμένα μέσω ορισμένων ανθρώπων που έκαναν κάποιες σκέψεις και που αρχικά είχαν πάρα πολλές δυσκολίες για να βρουν υποστήριξη για τις ιδέες τους. Συνεπώς λοιπόν η, η προσέγγιση ανταγωνισμός ε, για υπέρ της έρευνας νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω τον εισηγητή κοινή προσέγγιση, κοινή προβληματισμή και για τους δύο πυλώνες ε, έρευνα και καινοτομία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό πολιτικό μέλημα να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι ομιλητέ. Γι' αυτό κύριε Λαμπέρ, αν θέλετε να σχολιάσετε, έχετε τον ε, λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση αυτή. Νομίζω που ξεκίνησε, νομίζω θα πρέπει να συνεχίσει όταν υποβληθεί έκθεση. Αλλά νομίζω τα ζητήματα που ήγηραν οι συνάδελφοι βρίσκονται στο επίκεντρο τη συζήτηση. Δηλαδή, το να εξετάσουμε την εφαρμογή, την πρόκειται για μια έκθεση εφαρμογή. Το πλαίσιο υπάρχει και οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι, αλλά το ερώτημα είναι ε, κατά πόσο οδηγεί στην πρόοδο που επιθυμούμε όλοι μας από οικονομική, κοινωνική και οικολογική άποψη. Συνεπώς λοιπόν δεν υπάρχει κανένα, καμία, κανένα συγχωροχάρτη ε, για αυτή την παράληψη. Ε, λοιπόν, ας δούμε τι γίνεται στην Ήτρε. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, αυτή είναι η πρώτη φάση κίνησης των συζητήσεων και θα ενημερώσω του και συγητέ, γιατί για μένα είναι η πρώτη φορά μια τέτοια μορφή συνεργασίας μεταξύ δύο επιτροπών. Θα ενημερώσω λοιπόν τους Σικιώδης για την πρόοδο που σημειώθηκε και θα έχουμε την πλήρη συζήτηση στις 18 Μαρτίου στην Επιτροπή. Αλλά επιτρέψατε μου να πω το εξή. Νομίζω ότι μπορείτε να επενδύσετε πολλά ε, στην έρευνα αυτή καθευτή η έρευνα βασίζεται στην αριστεία παντού στον κόσμο. Εάν όχι, ε, μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό από τη βάση προς τα πάνω. Η καινοτομία στις διαδικασίες, η καινοτομία στις μορφές συνεργασίας. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη εμπειρία σχέση με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων Το θέμα είναι τι γίνεται για το, με το output των ερευνών αυτών, γιατί τις πολλούμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι μια θαυμάσια και ουσιαστική συζήτηση. Ας γίνει από κοινού λοιπόν με τις δύο επιτροπές. Εγώ όπως είπα θα σας ενημερώσω σχετικά και ίσως το καλοκαίρι θα ξέρουμε εάν είχαμε δίκιο να συνεργαστούμε με την Ήτρε ή όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λάμπερ. Νομίζω ότι πραγματικά σε θέση να δημιουργήσει αυτές τις ε, φιλίες με συναδέλφους από τις άλλες επιτροπές. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, δεν υπάρχουν άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να πω ότι συναφία με τους συνάδελφους συντονιστές θα κάνουμε την, ε, υπάρχουν, γραπτά υπάρχουν ορισμένα θέματα, θα γίνει συνεδρίαση. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι στα διάφορα, εγώ δεν έχω τίποτα να συζητήσω, εκτός αν κάποιος θέλει να θέσει ένα θέμα. Όχι, λοιπόν, τότε προσεχή συνεδρίαση, είναι βραχία συνεδρίαση, στις 22 Φεβρουαρίου, ε, μισή μέρα δηλαδή, από τις 3 έως τις 6.30,